Dear colleagues, dear commissioner. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε, ας ξεκινήσουμε. Yeah. No, no. The most important are here. Liebe Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφε. Ξέρω ότι θα έρθουν και οι υπόλοιποι, είμαστε λίγοι προς το παρόν, αλλά ε, δεν γίνεται να αλλάξουμε τρόπο διεξαγωγής συνεδρίασης τώρα το απόγευμα. Τηρώ χρονοδιάγραμμα και θα χτυπάω και το σφυράκι μου μέσα-μέσα γιατί ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και πρέπει να προχωρήσουμε όπως και το πρωί, αυστηρά. Ο εισηγητή λοιπόν θα κάνει μια παρουσίαση για 5 λεπτά, ο Σαλβαδόρ, μετά θα πάρει το λόγο ο επίτροπο και αργότερα η επίτροπο. Μετά θα, θα ακούσουμε μάλλον 10 λεπτά τον Επίτροπο και μετά θα πάμε στου εκπροσώπους των ομάδων οι οποίοι θα πάρουν το λόγο για 4 ή 5 λεπτά, θα δούμε. Έχω και κουδουνάκι εκτός από σφυράκι. Έχω διάφορα εργαλεία εδώ στη διάθεσή μου. Δεν θα το χρησιμοποιήσω όμως το, το κουδουνάκι γιατί έτσι ο, ο ήχος μου κάνει σαν να ήρθε ο Άγιος Βασίλης και ε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ επίκαιρο. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά μας, οπότε θα είμαι αυστηρή. Θα καλωσορίσω και πάλι εγκαρδίως τον Επίτροπο Κάλλας. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για, τους, για το δίκτυο μεταφορών στην Ευρώπη και θα παρακαλούσα τον εισηγητή να κάνει την πρώτη του παρέμβαση και μετά θα συνεχίσουμε όπως σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ από πλευράς μου τον Επίτροπο, διότι η Προεδρία, η Πρόεδρος συγκεκριμένα, είναι πολύ αυστηρή με το πρόγραμμά μας. Θα Συμμορφωθώ λοιπόν και εγώ αυτομάτως. Όπως ξέρετε οι μεταφορές είναι ένα τομέα που απασχολεί ένα εκατομμύρια ανθρώπου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι από τι πιο σημαντικέ μα πολιτικέ που ευθύνεται για ένα μεγάλο μέρο τη κατανάλωση και απορρόφηση και παραγωγή μάλλον του ΕΠ. Ε, μιλάμε για μια αγορά η οποία θέλουμε να είναι διέσιμη, βιώσιμη, ε, δημιουργεί θέσει απασχόληση και είναι μέρο τη στρατηγική μα και βεβαίω θα επηρεάσει και την αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών. Επίτροπε, βλέπουμε την πολιτική των μεταφορών ω ένα παράγοντα τη προστιθέμενη αξία του τομέα των μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν εδώ να αποφύγουμε την επικάλυψη που μπορεί να λαμβάνεται με δράσεις που μπορεί να σχεδιάζονται σε διεθνές επίπεδο και να περιορίσουμε τις δαπάνες. Θα θέλαμε λοιπόν την άποψη του Επιτρόπου, ε, την τοποθέτησή του για το ποιε επενδύσεις θεωρεί ότι θα πρέπει να καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο και ποιε σε κοινοτικό όταν μιλάμε για τις ε, δομές και τις υποδομές των μεταφορών. Χρειάζεται εδώ ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, διότι 4 δις ευρώ έχουν αποδοθεί από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα. Όσο έχουν τα πράγματα, υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης και επενδύσεων. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως να, γνωρίσουμε, να γνωρίζουμε το μέλλον των διευρωπαϊκών δικτύων. Όπω ξέρετε, Επίτροπε, το πρωί συζητήσαμε τι γίνεται με το φτωχότερο συγγενή των δικτύων αυτών, δηλαδή τα ενεργειακά δίκτυα. Τώρα ε, θέλουμε να περάσουμε σε αυτόν τον πλούσιο συγγενή ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ο Επίτροπος ίσως να μην τα θεωρεί τόσο πλούσια, όμως όσο έχουν τα πράγματα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών συγχρηματοδοτούνται λαμβάνουν ίδια ε, συνεισφορά από τα ΤΕΝ και από το Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής. Ε, θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε κατά πόσον θα βελτιωθεί η προστιθεμένη αξία τους. Και με έκθεσή μας για το θέμα αυτό γράψαμε ότι οι δαπάνες για το τομέα των του ΠΕΝ έφτασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ από το 1996 έως το 2020. Και παρόλα αυτά παραμένουν 500 δις τα οποία απομένουν να δαπανηθούν. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ταμείων και αύξηση της κοινοτικής συνεισφοράς στην κρηματοδότηση Τα δίκτυα αυτά δεν έλαβαν αρκετά κονδύλια στην τελευταία περίοδο προγραμματισμού, όπως είχε καταστήσει σαφέ ο εισηγητή του Κοινοβουλίου. Τι πιστεύει λοιπόν η Επιτροπή ότι θα πρέπει να γίνει για να σχεδιαστεί καλύτερα χρηματοδότηση των ΤΕΝ για τις μεταφορές. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης. Ξέρουμε όλοι ότι διαδραματίζουν εδώ ένα ρόλο οι εταιρικέ σχέσει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα πολλαπλά κριτήρια συμμόρφωση για να επιλέξει χρηματοδότηση. Χρειάζεται earmarking, δηλαδή εντοπισμό συγκεκριμένων ε, στοιχείων από τα ταμεία συνοχή και για το ερχόμενο διάστημα των δημοσιονομικών προοπτικών έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Η μία για το Γαλιλαίο, το πρόγραμμα αυτό, για το οποίο είναι σαφέ ότι στην κατηγορία 1α, με την οροφή που προβλέπετε, δεν έχει χρηματοδοτηθεί επαρκώ οι αναθεωρήσει και μεταρρυθμίσει ήταν απαραίτητε για να καλύψουμε αυτέ τι ελλείψει. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει επαρκή ευελιξία στι ισχύουσε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Και βεβαίω αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε συνεχώ κατά νου όταν θα σχεδιάσουμε τι ερχόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Εσεί τι νομίζετε, τι πιστεύετε για τον Γαλιλαίο. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα έπρεπε να κάνουμε ως προς τη χρηματοδότηση για τα ερχόμενα χρόνια και δεδομένων των αποτυχιών ε, που ε, ε, μας έφεραν οι σχέσεις, οι εταιρικές σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Τι θα γίνει στο μέλλον με αυτό και τι θα γίνει με το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Ουρανών, του European Skies. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τι αεροπορικέ μεταφορέ στο μέλλον. Ε, θα πρέπει να υπάρχει εδώ συνεπή χρηματοδότηση και απόδοση κονδυλίων συστηματικά για την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Επίτροπε, αυτέ ήταν οι βασικέ μέρημνε, τι οποίε θέλω να σα επισημάνω σε αυτή τη χρονική φάση και βεβαίω σημεία όπου θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε θέμενη αξία και εμεί ω Επιτροπή θα συνηγορήσουμε υπέρ του. Ήθελα λοιπόν να σας θυμίσω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε όθηση, νέα πνοή στον τομέα των μεταφορών, ε, τη ενέργειας και των επικοινωνιών ούτω ή άλλως. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τις δικές σας τι απόψει, Επίτροπε, διότι φαντάζομαι ότι και το κολέγιο των Επιτρόπων αυτά τα θέματα θα συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλο και βελτιώνεσαι, Σαββαντόρ. Θαυμάσια. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ε, άξι... Ε, χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω εδώ για τις μελλοντικές ανάγκες ε, των εξελίξεων στον τομέα των μεταφορών για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και όντως φτάνουμε σε ένα λεπτό πολύ σημαντικό που πρέπει να δούμε ε, τι θα κάνουμε διότι ε, ο, ο τομέας μας δεν είναι ένας μεγάλος τομέας Ευρωπαϊκής Ενώσεως για 10 δίκτυα ξοδεύουμε περίπου 1,1 ε, δις που είναι πολύ μικρό όχι μόνο σχετικά αλλά και σε απόλυτους αριθμούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, είναι μία πρόχειρη ε, μία πρόχειρη εκτίμηση διότι εδώ μιλάμε για 7 έτη δαπανών από τα διαρθρωτικά ταμεία και ε, για το Ταμείο Συνοχής για δαπάνες οι οποίες δεν απευθύνται μόνο σε μας και χρειάζεται να ε, συνεισφέρουμε και στην έρευνα και και ε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατά την περίοδο αυτή διότι οι μεταφορές σαν μέρος της υποδομής είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης οι ε, Ηνωμένε Πολιτείες και η Κίνα ε, ασχολούνται με πολύ μεγαλεπίβολα προγράμματα άρα εμείς πρέπει να την ανταγωνιστική μας θέση και θα πρέπει να μπορέσουμε να στηρίξουμε το, τα δικά μας θέματα διότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και υπολογίζουμε ότι ένα, ένα δισεκατομμύριο επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 18.000 θέσεων πέραν όμως αυτό υπάρχει αξιολόγηση ότι συνολικά θα έχουμε 1,2-3 εκατομμύρια και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ε, γιατί για να δημιουργήσουμε 10 δίκτυα ακόμη χρειαζόμαστε 500 δισεκατομμύρια δηλαδή θα υπάρχει χρηματοδότηση όχι μόνο από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα οπότε έχουμε ένα δίλημα αυτή τη στιγμή δηλαδή Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς ε, ετοιμάζουμε για τις ανάγκες τις μεταφορικές τον επόμενο, τον επόμενο χάρτη των των ε, διευρωπαϊκών δικτύων και προσπαθούμε να αναπτύξουμε την ε, έρευνα και την εξέλιξη ε, διότι για το μέλλον των μεταφορών ε, έχουμε ουσιαστικές προτεραιότητες ε, ουσιαστικά στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και συγχρόνως να διευκολύνουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί Ε, στον τομέα των ε, μεταφορικών δικτύων. Έχουμε ένα μεγάλο δίλημα. Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε επενδύσεις, άρα τι, τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε περιορισμούς ε, στον προϋπολογισμό, η κατάσταση είναι δύσκολη, και υπάρχει μία ατυχή στάση να καθυστερούμε και να αναβάλουμε τις μεγαλεπίβολες επενδύσεις και την υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων. Οπότε η Ευρώπη με τη σύγχρηματοδότηση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση των βασικότερων προγραμμάτων ε, για μεταφορικά δίκτυα. Ε, προς όχι μόνο μόνο της Ευρωπαϊκής αλλά και των κρατών μελών όπου θα εγκατασταθούν τα δίκτυα αυτά άρα θα πρέπει να υπάρξει και ένας κατάλογος προτεραιοτήτων ε, θα προσπαθήσουμε ε, να δούμε πώς θα υπάρξουν προγράμματα που θα είναι ε, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και γι' αυτό έχετε πολλά στοιχεία όπως άλλωστε το είπε και ο εισηγητής δηλαδή τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό διότι εφέτος το 2011 είναι ένα πολύ κρίσιμο έτος να δούμε αν προχωρά αρκετά γρήγορα το πρόγραμμα διότι διαφορετικά το κέντρο της Ευρώπης αν δεν διαχειριστούμε σωστά την κυκλοφορία θα έχει τόσους περιορισμούς ώστε δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα αναπτύξεως ούτε για τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές ούτε για γρήγορες αεροπορικές ε, ε, μετακινήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός που χρηματοδοτείται και είναι βασικό ότι έχουμε διάφορους ομολόγους που συμμετέχουν από πλευράς ιδιωτικού τομέα, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε όλους που έχουν τα κράτη-μέλη, άρα είναι βασικό να συνεχίσουμε αυτή την ε, ευγενή προσπάθεια. Σχετικά με τις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν. από τον εισηγητή. Ε, θα τις σκεφτώ κάπως. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινοτικό. και ε, θέλω να υπάρξει χρηματοδότηση ε, βέβαια για όλα τα προγράμματα που δεν είναι τόσο πολύ εύκολο για υπάρχει ε, ένας καυγάς για να υπήρξει ένας πυρήνας για τα μεταφορικά δίκτυα και υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και διαφορετικές δραστηριότητες περιφερειακές δεν είναι επίπεδο, ε, το πρόβλημα δεν είναι καν σε επίπεδο κρατών, είναι σε επίπεδο περιφερειακό και γι' αυτό εγώ θέλω να ε, προβώ σε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των υποχρεώσεων που θα είναι ευρωπαϊκές και αυτών που θα είναι εθνικές. Πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε να υπάρξουν αποφάσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κοιτάξει πώς θα τα προωθήσει. Ε, πρέπει να υπάρξει ένας πυρήνας που θα συζητηθεί και με το Κοινοβούλιο και το θέμα της ερεσιμότητος είναι πολύ σημαντικό και αντικρουόμενο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με, ε, πολύ ευχάριστα με την Γενική Διεύθυνση ε, Ρέτζιο κατά τρόπον ώστε να υπάρχει σωστή χρήση των ε, διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής διότι διαφορετικά πώς θα μπορέσουμε μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει στην πρακτική βέβαια, αλλά πρέπει να υπάρχει μία προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή διασυνοριακή και ε, να υπάρξει και συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ήδη ότι η συνοχή αυτή στον ε, τομέα αυτό θα αντιμετωπίσει μεγάλη αντίσταση από πολλά κράτη-μέλη και γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες των συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να καθορίσουμε τις δυνατότητές μας σε, από πλευράς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και θα δούμε πώς μπορούμε να εμπλέξουμε και τα ιδιωτικά κεφάλαια αλλά τώρα τέλειωσε η ώρα μου άρα τέλειωσε. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τη σειρά των των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων θα λάβουν το λόγο. Καταρχήν για το ΕΛΚ, ο Μαριζό Μαρινέσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύων είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Έχουμε πολλά project τα οποία τρέχουν σε διάφορε ε, περιοχές και είναι και σε διάφορες φάσεις της εφαρμογή τους. Βέβαια η ε, κατανομή των κονδυλίων δεν ήταν επαρκής, εξαρτιόταν από το Ταμείο ε, Συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης δεν υπήρξε πολύ καλό συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης ε, συμπεριλαμβανομένου και του εθνικού προπολογισμού. Οπότε μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτών των προγραμμάτων ολοκληρώθηκε. Τώρα η Κομισιόν κάνει διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη ώστε να επαναπροσδιορίσει τις δομές και τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν να τεθούν κάποιε βασικές αρχές ώστε να υπάρξει επιπλέον προστιθέμενη αξία να ορίσουμε ας πούμε κάποια προγράμματα προτεραιότητας ε, επί τη βάση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που αυτά θα επιφέρουν. Ε, Οι στρατηγικοί ευρωπαϊκοί άξονες από, ε, από, των διεξόδων όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για... και πρέπει να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά που θα μπουν σε αυτές τις ε, κατηγορίες. Συντονισμός των προγραμμάτων που, που ε, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, ε, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς προπολογισμούς, ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές επιρροές που, έχει... που έχουν τα προγράμματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να δούμε Πώ θα συμβάλλουν και τα κράτη-μέλη σε όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να κεφαλοποιήσουν στις υποδομές τους. Επίσης έχουμε το πρόγραμμα της ανταλλαγής εκπομπών αερίων. Έχουμε και την Ευρωβινιέτα. η συμπερίληψη επίση τη ε, συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, η προώθηση των ΣΔΙΤ. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη υποστήριξη έτσι ώστε στι ε, μελλοντικέ οικονομικέ προοπτικέ να υπάρχει μεγαλύτερο ποσό για τα ευρωπαϊκά δίκτυα από ό,τι υπάρχει τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η δική μου πολιτική ομάδα σας θεωρεί ως κάποιον που θέλει να υπάρξει πρόοδος στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ό,τι είπατε αντικατοπτρίζει και τις δικές μας προσδοκίες και είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε λίγο την προοπτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξουν πιο πολλές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τώρα μόνο τα εθνικά κοινοβούλια, είναι αυτά, ε, τα, εθνικά, τα κράτη-μέλη μάλλον είναι αυτά που συμβάλλουν περισσότερο. τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, ε χωρίζονται σε τομείς στα διάφορα κράτη-μέλη και ναι, όντω έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχει ανάγκη για σωστή επαρκή χρηματοδότηση. Αυτή είναι και μία από τι βασικότερε προκλήσει. Όλε οι, πηγέ οι πηγές χρηματοδότησης θα πρέπει ίσω να γίνουν μία. διαρθρωτικά ταμεία δηλαδή, ταμείο συνοχή, ε, κονδύλια που έχουν αποδοθεί στα, στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ίσως θα πρέπει να, τα, να, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας ώστε να γίνεται καλύτερη κατανομή αυτών των ε, κονδυλίων. Βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη και η, ε, η Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και τα ΣΔΙΤ. Βεβαίως υποστηρίζουμε την διαφοροποίηση των πηγών αν αυτό σημαίνει περισσότερα κονδύλια και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι και έχετε σκεφτεί αυτό ήδη. Τώρα, προτεραιότητες. Ε, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητε, υποστηρίζουμε την προσέγγιση του δικτύου. Ας προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε διάφορους τομεί σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά κενά αυτή τη στιγμή. Εγώ εκπροσωπώ ένα νέο κράτος μέλος και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το δίκτυο το σιδηροδρομικό έχει, το έχουμε ξεχάσει. Στη δική μου χώρα μόλις 10% του προϋπολογισμού πάει στους σιδηροδρόμους. Το υπόλοιπο 90% πάει στις οδικές μεταφορές. Είναι ξεχασμένο λοιπόν αυτό το δίκτυο και νομίζω ότι αυτή η πρακτική θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα για τις μικρότερες προτεραιότητες νομίζω ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την γεωγραφία και σε ό,τι αφορά τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό είναι μια βασική ιδέα Γιούτα, αν ε, ε, μίλησα πολύ, αν πέρασε ο χρόνος μου, χτύπα το σφυράκι σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, αυτά ήθελα, Πρόεδρε, να πω για το, στον Επίτροπο. Ε, είπα δεν θα κουνάω το κουδουνάκι γιατί δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης που έρχεται με τα δώρα θα χτυπάω το σφυράκι μου όμως αν χρειαστεί εντάξει νομίζω ότι δεν ξεπέρασε τον χρόνο σου μην ανησυχείς η κυρία Γένσεν έχει το λόγο. Ε, είναι αξιέπαινε οι προσδοκίε που έχετε κύριε Επίτροπε για τον τομέα των μεταφορών και ελπίζω ότι θα, να, θα μπορέσει και το Κοινοβούλιο να σα στηρίξει. Ε, ένα απλό ερώτημα ήθελα εγώ να θέσω η κατάσταση ποια είναι, πού είναι το, πού είναι το πρόβλημα. Δεν έχετε χρήματα για τα, από τα διευθυντικά ταμεία για τις μεταφορές, δεν έχετε χρήματα για, την, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και τι γίνεται με τα 30 προγράμματα προτεραιότητας. Τι μπορεί να γίνει. Πού, πόσο μακριά είμαστε από το να επιτύχουμε τους στόχους μας εφόσον έχουμε βρεθεί σε, αυτή την, ε, σε αυτό το διέξοδο και πού χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αυτό το που είπε και ο κύριος Λιμπεράτσκι, το θέμα της ε, δημιουργίας ενός ταμείου μεταφορών ώστε να υπάρχουν ε, αυτοτελή κονδύλια εκεί Ίσως αυτό να πρέπει να είναι, γιατί ε, ούτω ή άλλω ένα κομμάτι των κονδυλίων από τα διευθυντικά ταμεία πάει στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό να περάσει και από το Συμβούλιο, ακόμη και εδώ στο Κοινοβούλιο θα είναι δύσκολε οι συζητήσει. Η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο δεν το επικροτεί ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Υπάρχουν και εδώ διαφορετικέ απόψει. Ξέρω ότι ε, θέλετε, τι θέλετε να πετύχετε, αλλά πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτή, να ξεπεράσουμε αυτή την αντίσταση που υπάρχει για τα, από τα κράτη-μέλη που θέλουν να διατηρήσουν το δικό του σχεδιασμό και ταυτόχρονα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να κατασκευαστούν και τα δίκτυα. Και κάτι τελευταίο. Ποια είναι η άποψή σα για τα μικρότερα προγράμματα. Όχι για τα βασικά δίκτυα, αλλά και για μικρότερα δίκτυα, όπου έχουμε στα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα προγράμματα σήμερα ε, με αιτήσια συνεισφορά. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα καλά προγράμματα, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για όλα αυτά τα προγράμματα. Σω λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν και διευρωπαϊκέ λύσει ή πιο αποτελεσματικέ μεταφορέ, καλύτερε λύσει που να λαμβάνουν υπόψη και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, ε, εξοικονόμηση ενέργειας, ε, να φύγουν οι μεταφορέ αποκλειστικά από, το, από την οδική αρτηρία που βρίσκονται τώρα. Ίσως λοιπόν και τέτοια προγράμματα θα χρειάζονταν χρηματοδότηση. Η δική σας άποψη ποια είναι για αυτά τα μικρότερα ε, ίσονος ίσως σημασίας ε, προγράμματα των διευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Ιζαμπέλ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά σχόλια, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τη συζήτηση αυτή από το τι γίνεται με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο στι μεταφορέ και από την άλλη με τη λευκή βιβλίο που περιμένουμε, από την Επιτροπή, περιμένουμε στην Επιτροπή Μεταφορών και ε, με του ιδίου πόρου. Το θέμα του αν θα αποδώσουμε στον τομέα των μεταφορών Ό,τι προσπαθούμε να ξαναπάρουμε από τη δασμολόγηση των υποδομών λόγω χάρη, αυτό είναι ένας κίνδυνος. Αναποκλειστικά τα πάμε όλα εκεί διότι μπορεί όχι απλώς να εσωτερικεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα εξωτερικά κόστη και να τα καλύψουμε, αλλά να προκαλέσουμε και πολλές κινδύνους και έλλειψη ισορροπίας. Δεν ε, πρέπει να γίνουν όλα στον τομέα των μεταφορών έτσι απότομα. Επίσης, τα στοιχεία στοιχείο κλειδί είναι η κατανομή των δικτύων μεταξύ διευρωπαϊκών δικτύων και συνοχής ε, για παρόμοια δίκτυα όπως τα οδικά. Οι αριθμοί νομίζω είναι εύκολο ότι το γνωρίζετε και Πρέπει να δούμε την ποιότητα των κριτηρίων επιλεξιμότητα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα ταμεία συνοχή. Αλλά κυρίω την συνοχή, τη συνεκτικότητα εδώ. Μιλάμε για συντονισμό. Ποια όμω η συνέπεια μεταξύ ορισμένων επενδύσεων στα διευρωπαϊκά δίκτυα από τη μια και από την άλλη των όσων κάνουμε ή δεν κάνουμε από την πλευρά τη συνοχή, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη νομοθεσία για το περιβάλλον, τη χωροταξία σε περιφερειακό επίπεδο. Εκεί τι γίνεται με το συντονισμό Μιλάμε για πραγματικά, πραγματική λήψη συνέπειας. Ορισμένα μεγάλα έργα οδικά είναι τελείως ε, αντιφατικά με όσα θέλουμε να κάνουμε σε άλλου τομεί. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον. Και επίση ξέρουμε ότι στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κάτι μέλη που πάντοτε δίνουν ε, μεγαλύτερη σημασία στα εθνικά του δίκτυα και όχι τα διασυνοριακά τα διακρατικά και εμείς ξέρουμε ότι εδώ επιδιώκουμε το διακρατικό και κάνουν επενδύσεις στα συνδυοδρομικά τους δίκτυα που τους επιτρέπουν να ε, κάνουν εξοικονομήσεις για το μέλλον. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, εάν στο RTMS ε, επίτροπε επενδύσουμε περισσότερο ένα νέο σύστημα για τους σιδηροδρόμους θα ε, κερδίσουμε για το μέλλον, διότι θα επιτρέψουμε να κερδίσουν κάποιοι με τους επιπλέον φόρους που επιβάλλονται και μετά να επενδύσουν στην βελτίωση των υποδομών. Θέλουμε λοιπόν ναι να δράσουμε γρήγορα, αλλά όχι με περιττές δαπάνες είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Και για, συνέπεια, για λόγω συνέπειας να σκεφτούμε και τα κονδύλια της έρευνας ε, με το πρόγραμμα αυτό που όλοι γνωρίζετε καλά, το ITER για το 2020, αλλά και το πρόγραμμα Galileo, το οποίο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το ITER το ίδιο. Διότι αν κάνουμε σύγκριση μεταξύ της στρατηγικής ε, ε, ένταξης του προγράμματος αυτού σε γεωγραφικό επίπεδο και το πώ μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέε τεχνολογίε. Σκεφτείτε τι μπορείτε να εξοικονομήσετε με τον Καλιλαίο, το GPS, τα νέα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται θα αποφύγουμε ε, το να διανύουμε χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων ε, άδικα, εισμάτιν. Εδώ ε, πρέπει να σκεφτούμε και τους σκοπούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. ECR, ο κύριος Φάιμον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η δική μου ομάδα θεωρεί ότι το πιο σημαντικό είναι το ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία. Και ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι αυτά τα οποία μπορούν να έχουν αυτή τη μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ναι, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Η... Τα ευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να τα δούμε προσεκτικά και τους ε, σιδηροδρόμους και, τους, ε, και τις οδικές αρτηρίες. Θα δείτε όμως ότι αν τα δούμε όλα αυτά υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ κεντρικής, ε, δυτικής, ανατολικής Ευρώπης. Η κεντρική Ευρώπη δεν είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την δυτική Ευρώπη και εδώ υπάρχει τεράστιο δυναμικό για επιπλέον προστιθέμενη αξία για την ε, καλύτερη δηλαδή ε, σύνδεση των ε, κεντρικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Δυτική ή ας πούμε ή με τις χώρες της Βαλτικής. Οι χώρες της Βαλτικής δεν συνδέονται εξαιρετικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και το ίδιο ισχύει και για τις βαλκανικές χώρες. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση εσείς, θεωρείτε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ δεν βλέπω κανέναν. Από την EFT επίσης δεν βλέπω κανέναν. Οπότε πάμε... Α, όχι, όχι, όχι. Λάθος, λάθος. Έχουμε την μεγάλη τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών μαζί μας. Έχουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, παρακαλώ, Μπράιαν. έχεις το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μένα είναι αλλαγή να κάθομαι από αυτή τη μεριά και όχι από τη δική σας στο Προεδρείο. Εδώ Ακούσαμε να προβάλλονται επιχειρήματα υπέρ της πολιτικής μεταφορών. Ακούσαμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή κάποια επιχειρήματα, αλλά όταν έφτασε είδα πολλά οικεία πρόσωπα είναι σημαντικό λοιπόν ότι μας καλέσατε στην Επιτροπή σας. Είναι επίσης σημαντικό ότι διοργανώσετε σήμερα αυτή τη συζήτηση καθώς και η παρουσία του Επιτρόπου είναι εξίσου σημαντική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σήμερα το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετό χρήμα, αρκετά κονδύλια για να φτιάξουμε όσα επιδιώκουμε. Πρέπει λοιπόν να αποσπάσουμε όλη όσο περισσότερη προστιθέμενη αξία μπορούμε από τα κονδύλια που διατίθενται. Είναι νομίζω σημαντικό για μας τις μεταφορές να μπορέσουμε να δώσουμε οι ίδιοι μια προοπτική στις μεταφορές. Να σκεφτούμε τι μπορεί να προσφέρουν οι μεταφορές στην στρατηγική του 2020, στην ανάκαμψη της εργασίας, της απασχόλησης, στη βιωσιμότητα. Όχι τι θέλουν οι μεταφορές να πάρουν από, τα άλλα, από τους άλλους τομείς. Εάν σκεφτούμε λοιπόν αυτό αυτή, αυτό το εγχείρημα που είναι και πολιτικό και όχι απλώς από την άποψη των εκτιμάτων και μειονεκτημάτων, θα πρέπει να δούμε ότι στην οικονομική ανάκαμψη και στη στρατηγική αυτή οι μεταφορές είναι καθοριστικός παράγοντας. Είναι καθοριστικός παράγοντας στη συνολική σύλληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη κυκλοφορία μεταφορών και ανθρώπων, και, ανθρώπων εμπορευμάτων και πολιτών. Χωρίς μεταφορές δεν μπορεί να, μετακινηθούν τα εμπορεύματα. Ούτε μπορεί να προκύψει οικονομική ανανέωση. Για μας λοιπόν ως Επιτροπή Μεταφορών είναι σημαντικό να σα διαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα σε εσά και του συναδέλφου σα καθώ επιτελείτε το έργο σα. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να διαδοθεί ευρέω. Όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο και σε όλα τα θεσμικά όργανα. Υπ' αυτήν την έννοια Είναι σαν να μιλάμε για, το, για ήρωες από western ε, όταν μιλάμε για τους υπεύθυνους των μεταφορών που θέλουν να σας πάρουν ε, με την απειλή περιστρόφου τα χρήματά σας. Όχι. Θέλουμε την καλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για τις μεταφορές από τις υπάρχουσες δημοσιονομικές γραμμές και να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους ή δυνατόν για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Τις παρατηρήσεις τις έχουν κάνει ήδη συνάδελφοι από την Επιτροπή Μεταφορών. Πρέπει όμως και εγώ να σταθώ στα εξή. Πρώτον, πιστεύουμε στην Επιτροπή Μεταφορών ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Οι ημέρες των 27 εθνικών μεταφορικών πολιτικών που ισχύουν ταυτόχρονα ώστε να μιλάμε τελικά για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με κάποια συγκεκριμένα σημεία περάσματος στα σύνορα πρέπει να ξεπεραστεί. Είναι σημαντικότατος ο παράγοντας ο διασυνοριακός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το, η ταχεία από τη Μαδρίτη στη Βαρκελόνη η οποία φτάνει στο Περπινιάν. Όμως δεν υπάρχει σύνδεση Βαρκελόνης με Περπινιάν. Άρα αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει μαζί να περάσουμε τα σύνορα, να τα διαβούμε και να διασυνδέσουμε τα εθνικά συστήματα προκειμένου να προωθήσουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό θα είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Επιπλέον, Πρόεδρε, εάν η αηφορία είναι σημαντική, σκεφτείτε το εξής. Εάν θέλουμε ε, βιώσιμο μεταφορικό δίκτυο, αυτό θα ωφελήσει και το περιβάλλον και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Δεν μιλάμε εδώ απλώς για στρώσιμο σιδηροδρόμων ή για να στρώνουμε άσφαλτο τυχαία. Όχι. Και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και για την αύξηση των κονδυλίων που θα αφιερωθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και βάσει της στρατηγικής του 2020. Σήμερα άκουσα τον ε, Βρετανό Υπουργό μετά από διάσκεψη στη Βουλή των Λόρδων να λέει ότι πρέπει να λάβει περισσότερα χρηματοδοτήσεις στη Μεγάλη Βρετανία για τα δίκτυά της από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όμω δεν πάνε έτσι τα πράγματα και κάποιο να το πει αυτό στο Βρετανό Υπουργό. Έτσι. Λοιπόν, για τα μεγάλα έργα υποδομών χρειάζεται σίγουρα κάποια αύξηση, αλλά είναι τεράστια και η απόσταση μεταξύ του τι χρειαζόμαστε και το τι έχουμε διαθέσιμο για δαπάνη αυξημένο συντονισμό μεταξύ των υπαρχόντων ταμείων, των ε, διευρωπαϊκών δικτύων δηλαδή και ε, των ταμείων Συνοχή. 23% των δαπανών τη συνοχή, Πρόεδρε, γίνεται για τι μεταφορέ. Όμως, όταν δαπανεί κανείς τα κονδύλια της συνοχής, σκέφτεται τις μεταφορικές πολιτικές, τις προτεραιότητες των μεταφορών που απαιτεί και χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν δείτε τους αριθμούς, Υπάρχουν τεράστια ποσά που θα για τα οδικά δίκτυα χωρίς να είναι αυτοπροτεραιότητα ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάμε για μετακινήσεις, για μεταφορές. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει στενότερος σχετισμός των προτεραιοτήτων των μεταφορών με, τις, με τη συνοχή και τις δαπάνες που γίνονται από το Δομείο Συνοχής. Τέλος, Πρόεδρε, να πω το εξής ενδιαφερόμαστε για όλα αυτά τα ζητήματα και πιστεύουμε συνεχώς ότι θα βρούμε κάποια λύση. Ο κ. Μπαρόζο όποτε του ζητάω ένα... Όταν μιλάμε για λύσεις στα προβλήματα που αναζητούμε και το αναφέρω όλα αυτά που μας απασχολούν, μου βρίσκει μια μαγική λύση, μια μαγική συνταγή. Τα ομόλογα. Εδώ χρειαζόμαστε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, για τις εταιρικές σχέσεις δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Στο παρελθόν δεν υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχίες. Γιατί, Γιατί το κοινό το κομμάτι μάλλον του δημόσιου τομέα να λαμβάνει όλο τον κίνδυνο, ενώ ο ιδιώτης όλο το κέρδος. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να εξακολουθήσει. Χρειαζόμαστε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης για τις μεταφορές. Και κάποιοι μίλησαν και για το λεγόμενο, ε, για την περιχαράκωση κάποιων κονδυλίων. Ένας όρος που χρησιμοποίησε και ο Βρετανός Υπουργός που σας έλεγα, το ring fencing αυτό όσοι το επιχείρησαν απέτυχαν και στα 27 κράτη-μέλη. Όμως είναι και αυτός ένας τρόπος χρηματοδότησης. Είναι ένας τρόπος να ε, σκεφτεί κανείς τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Και κάτι άλλο που θα θέλει να προωθήσει η Επιτροπή μας προς τη δική σας είναι το εξής. Εάν τα κράτη-μέλη λαμβάνουν κονδύλια από την Ευρώπη και δεν τα χρησιμοποιούν, να τα χάνουν όχι να πηγαίνουν στα εθνικά θησαυροφυλάκια αλλά πίσω στα ευρωπαϊκά ταμεία, όπου μπορούν να αξιοποιηθούν για σημαντικά έργα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τον χρόνο σας και ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρέμβω. Ευχαριστώ. Ε, είναι ένας ε, πρέσβης ο κύριος Σίμψον ε, των μεταφορών. Καλύτερο πρεσβευτή των ιδεών της Επιτροπής Μεταφορών δεν θα μπορούσατε να έχετε βρει. Έχουμε 6-7 άτομα στον κατάλογο. Τσέλερ, Οντί, Κρέλ, Βον, Πίπερ. Κλείνω εδώ τον κατάλογο και θα πάρετε το λόγο ο καθής για δύο λεπτά. Και μετά κύριε Επίτροπε έχετε εσείς το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος Σίμψον έθεσε τα βασικά σημεία για την Επιτροπή, ε, της Επιτροπής Μεταφορών, μας τα παρουσίασε και μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε. Ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ξεπεράσει τα σύνορα. Και ένα από τα θέματα που προωθούμε είναι η κινητικότητα. Προφανώς σε αυτό ε, πρέπει να ξεπερασει τα συνορα και ενα απο τα θεματα που προωθουμε ειναι η κινητικοτητα προφανως αυτο πρεπει να ενταχθει και το θέμα ε, των μεταφορών για να μπορέσουμε να, να διαχειριστούμε τις ροές ατόμων και ε, αγαθών ε, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε δύο σημεία για τις, ε, για τις μεταφορές, εντάξει υπάρχουν κάποια προβλήματα, καταρχάς το θέμα των ε, αεροπορικών μεταφορών με το Single European Sky και οι συνδρομικές μεταφορές. Όταν η μεγαλύτερη εταιρεία επιμελητία στην Γερμανία λέει ότι 60% των ε, αγαθών ε, γίνονται με, αεροπορικά, ε, με αεροπορικές μεταφορές και 40% στο δρόμο, οδικά και σιδηροδρομικά, τότε προφανώ οι σιδηρόδρομοι δεν παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί δεν είναι τόσο ευέλικτοι. Οπότε τόσο ευέλικτο αυτό ο τομέα μεταφορών. Απ' την άλλη, όταν οι αποστολείς θέλουν να επιτρέπονται τα gigaliners που λέγονται στην, ε, στους δρόμους, ε, προφανώς αυτό χρειάζεται και κατάλληλη ε, υποδομή. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που θέλουμε να κυνηγήσουμε με την ε, πολιτική για το 2020. Αν λοιπόν θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά, πρέπει να τα δούμε στα μάτια. Ναι, διευρωπαϊκά δίκτυα και τα υπόλοιπα ε, βήματα θα πρέπει να το δούνε και σημαντικά και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώ γίνεται τελικά. Τι θα κάνουμε. Ε, δημόσια χρηματοδότηση. Εντάξει, ναι, αλλά το 1 τέταρτο της, των κονδυλίων από τα διερθωτικά ταμεία και από τη συνοχή πάει στα, στις μεταφορές. Την επόμενη λοιπόν ε, περίοδο ε, θα πρέπει να περιγράψουμε πού ακριβώς θα πρέπει να πάνε τα κονδύλια, από πού θα πρέπει να φύγουν, πρέπει να δώσουμε μια κατεύθυνση. Για να μην παραμείνουν όλα αυτά όνειρα θερινής νυχτός. Και ναι, οι προπολογισμοί των κρατών μελών δεν ε, κατανέμουν συγκεκριμένα ποσά πάντα στοχοθετημένα αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουν οι, τα, ε, τα κονδύλια αυτά να εισρέψουν στον τομέα των μεταφορών για να μπορέσουν και οι μεταφορές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε τα ΣΔΙΤ, δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε τα πράγματα μόνο από το δημόσιο τομέα. Νομίζω ότι αυτά ακόμη έχουν παραμείνει εκκρεμή και πρέπει να τα λύσουμε. Ευχαριστώ ε, κύριε Τσέλερ. Ο κύριος Ροντή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω, ε, ε, θέλω να σας έχω εμπιστοσύνη κύριε Επίτροπε. Είστε ένα σοβαρό άτομο. Όταν ήσασταν ο, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Εστονίας είστε, είχατε γίνει ο πατέρας της κορώνας της Εστονίας και έχω λόγο να σας εμπιστευτώ. Πρέπει να επενδύσουμε όχι όμως μόνο στις μεταφορές, στην, ε, ναι, στην ε, στο, στην ψηφιακή τεχνολογία, στο νερό. Έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεω και ε, θέτω όλα αυτά τα θέματα προ συζήτηση και στην Επιτροπή σας κυρία Πρόεδρε, διότι τώρα πρέπει να, στη συζήτηση για τον προπολογισμό να έχουμε ένα τμήμα ε, σχετικό με τις επενδύσεις για να μπορούμε να ε, χρηματοδοτήσουμε πολύ διετής ε, επενδύσεις πέραν της εφταετίας. Δεύτερον, όσον αφορά τους πόρους και τα μέσα, πρέπει να δούμε αν δεν πρέπει σε συνεργασία με τους εθνικούς βουλευτές να κάνουμε έναν λογιστικό έλεγχο της, της ε, διαδικασίας μεταξύ κράτους περιφερειακών αρχών και τοπικής αυτοδιοίκησης διότι μας λέγεται ότι μπορούμε να κάνουμε κάνουμε πολύ, ε, πολλές οικονομίες. Έχουμε 27 στρατούς και συν μία το, την κεντρική 28. Πάρα πολλά διπλωματικά κτίρια σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με τις Εθνικές Ελεκτικές ε, Αρχές να κάνει αυτό τον έλεγχο και θα μπορέσει μπορέσουμε να ε, αποδεσμεύσουμε έτσι σημαντικούς πόρους οι οποίοι θα μπορούν να αφιερωθούν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στην ε, ε, ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η κυρία Κρέλ η πολιτική συνοχής δεν είναι πολιτική μεταφορών και φαντάζομαι ότι σε αυτό το σημείο συμφωνούμε όλοι. Αλλά η περιφερειακή εξέλιξη χωρίς μια λογική πολιτική δεν είναι εφικτή. Γι' αυτό και πρέπει και στο μέλλον, στον τομέα της, της ε, πολιτικής συνοχής να ε, φροντίσουμε για μια ε, λογική ρύθμιση των μεταφορών. Επιζητούμε προστιθέμενη αξία. Συμφωνώ με τον Brian Simpson που που λέει ότι οι δυνασιονοριακές επικοινωνίες είναι σημαντικές και πρέπει να προωθηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και δύο άλλα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε δηλαδή ποιος είναι ο λόγος να δεσμεύουμε ε, για προγράμματα μεταφορικά σε κάποιο κράτος πόρους όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Ισπανίας και Γαλλίας και δεν συμβαίνει τίποτα. Έχουμε δεσμευμένα εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορούν να δοθούν, να επιστραφούν στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο. Αυτοί οι πόροι μπορούν να επιτρέψουν να εφαρμόσουμε μια διαφορετική πολιτική μεταφορική. Επίσης ε, είπαμε ότι εμείς ψηφίσαμε την ε, γνωμοδότησή μας στην Περιφερειακή Επιτροπή και ζητήσαμε ε, σαφώς να μην επιστρέφονται τα ποσά του, πόρου, του Ταμείου Συνοχής στα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μπορούν να παραμείνουν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα είναι μεγάλη μάχη, αλλά θα μπορούσαν τότε να χρησιμοποιηθούν και για προγράμματα μεταφορών. Ευχαριστώ. Ο Ντέρεκ έχει το λόγο. Μια γενική παρατήρωση, παρατήρηση Πρόεδρε, και έπειτα μια ερώτηση προς τον Επίτροπο. Κάτι που έθιξε και ο ίδιος στην παρουσίασή του. Η γενική παρατήρηση μου ήταν μετά την παρέμβαση του συναδέλφου του κυρίου Σίμψεν. Ο Μπράιαν ο συνήθως ε, ήταν ε, ενθουσιώδης υπέρ της μεταφοράς, της πολιτικής μεταφορών και έχει δίκιο. Διότι για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται συντονισμός με τόσο μεγάλα έργα υποδομών για τις μεταφορές που προβλέπονται. Πρέπει όμως για το μέλλον να προβλέψουμε και χρηματοδότηση είτε μέσω των ομολόγων, είτε μέσω του Ταμείου Συνοχής είτε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από, από, επενδύσεων, από όπου και να έρθουν τα κονδύλια, πρέπει να τα εξεύρουμε γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε και του συσχετισμού των μεταφορικών δικτύων, αλλά να δημιουργήσουμε και θέσει εργασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το συγκεκριμένο ερώτημα που έχω προ τον Επίτροπο αφορά το σχέδιο, το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ, που ανέφερε στην παρουσίασή του. Όταν μίλησα στην βιομηχανία που ασχολείται με τα θέματα αυτά πρόσφατα, θεώρησαν ότι εδώ μπορεί να μην είμαστε αρκετά γρήγοροι και να μας προλάβουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί καθυστερούμε. Μπορεί να μας πει εάν θεωρεί και εκείνο ότι κάπως δεν έχουν τα πράγματα, μπορεί να μας προλάβουν οι Ηνωμένε Πολιτείε το πρόγραμμα αυτό. Πίπερ. Ο Μάρκος Πίπερ. Yeah, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και εγώ προέρχομαι από την ε, Επιτροπή Περιφερειών και αντιλαμβάνεστε ότι ε, εκεί αναγνωρίζεται η προστιθέμενη αξία των μεταφορικών δικτύων, γι' αυτό και θα θέλαμε ε, να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται προτού εφαρμοστούν ορισμένα αξιέπαινα προγράμματα, αλλά αυτό το οποίο δεν θέλουμε θέλουμε να υπάρξει είναι ένα ταμείο μεταφορών διότι τότε θα ε, συγκεντρωθεί ε, στην Ευρώπη ε, μία ευθύνη και θα ήθελα να ξέρω τι μπορείτε εσείς να μας εξασφαλίσετε και πώς μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι μία τέτοια κεντρική δακτηριότητα δεν θα καταλήξει σε μία απλώς θέση των ε, περιφερειών που θα πληρώνουν αλλά δεν θα συμμετέχουν. Λοιπόν, ε, ε, ευχαρίστως να συμμετάσχουμε εις τα δίκτυα, θα συμφωνήσουμε, αλλά πέραν αυτού τα χρήματα είναι δαπανηρά και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποδοτικά. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε αν δεν θα πρέπει να επενδύουμε όπου υπάρχει ήδη μεγάλη κίνηση, μεγάλη κυκλοφορία διότι αν εκεί υπάρχουν κενά, υπάρχουν αδιέξοδα, ε, αν υπάρχει συμφόρηση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο εποφελώς η χρηματοδότηση από την δημιουργία ενός νέου αυτοκινητοδρόμου από το μηδέν. Ευχαριστώ. Είναι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να εκφράσω την ικανοποίησή μου που εξετάζουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Και το θέμα των μεταφορών και τον προπολογισμό που θα του αποδοθεί. Ευχαριστώ λοιπόν και εσά, Πρόεδρε, και τον Επίτροπο για την παρουσία του σήμερα το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα, ένα σύντομο σχόλιο για το γεγονό ότι διαρκώ το λέμε και μάλιστα και πριν από τα Χριστούγεννα ότι η Σιδηρόδρομη είναι πολύ σημαντική. Ο Γάλλος και ο Ισπανός υπουργό συζητούν τα θέματα αυτά και ελπίζουμε ότι στον Δεκέμβριο θα καταφέρουμε να λειτουργήσει πλέον αυτή η σύνδεση Περπινιάν Βαρκελόνης. Βεβαίως, το να υπάρχει κεντρική διαχείριση μας προκαλεί ανησυχίες και το πρόβλημα είναι κατά πόσον η χρηματοδότηση της Ισπανίας ε, συμμορφώνεται με τις, υποχρεώσεις χρηματοδότησης που προβλέπονται ή σε περιφερειακό επίπεδο οι υποδομές που απαιτούνται τελικά δεν πραγματοποιούνται, δεν ε, χτίζονται. Εδώ λοιπόν ζητούμε από την Επιτροπή να πιέσει τα κρατη να καταφέρουν να δουν ότι υπάρχει σε μερισμένα πράγματα ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία από το να επιμένουν στα δικά τους εθνικά συμφέροντα και μόνον. Ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πιστεύετε ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να δείξει την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προσπαθειών, του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτό σε πολλούς τομείς πολιτικής, ε, κύριε Επίτροπε, όπως την έρευνα, τις τεχνολογίες, τα διευθυντικά ταμεία, τη γεωργία, εκεί θα θέλαμε η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να είναι κάτι στο οποίο θα δοθεί έμφαση, να γίνει κάτι που θα καταστεί σαφές όταν μιλάμε για τη διασυνοριακή διάσταση. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, πρέπει να είναι κάτι που θα υπογραμμίζεται διαρκώ. Πέρα από τη συνοχή, την κοινωνική, εδαφική, οικονομική συνοχή. Πώς πιστεύετε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μπορούν να συνεισφέρουν στο, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής το 2020 και να εξυπηρετήσουν την ε, ευρωπαϊκή μηχανία. Για μας είναι σημαντικό να επενδύσουμε στις υποδομές, όχι μόνο στους σιδηροδρόμους, όχι μόνο στους αυτοκινητοδρόμους, αλλά για την ίδια τη βιομηχανία είναι σημαντικό. Θέλουμε κάτι παρόμοιο να συμβεί και εδώ. Ε, και τέλος, ο κύριος ο κύριος Λαμασούρ που δεν είναι εδώ τώρα, όλοι ξέρουν ε, για τα θέματα συνοχής πόσο έχουμε προβληματιστεί. Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα με ευρωμόλογα. Ευχαριστούμε Τα κατέστρεψε όλα όσα έχτισα για την ε, πειθαρχία στο χρονοδιάγραμμα, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Ένα ερώτημα, Πρόεδρε, για τον Επίτροπο. Όταν πήραμε τον προπολογισμό για το 2011, προτείνεται 10% αύξηση για την υποστήριξη των ε, διεθνών ε, δικτύων. 725 εκατομμύρια δηλαδή. Από 725 εκατομμύρια σε 810. Ε, στο, εμείς σας υποστηρίξαμε, αλλά το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο δεν το ε, υποστήριξε. Άρα αφαιρέσαμε 2,3%. Είχαμε το Μαρκοπόλο 49%, ε, το Τσέζαρε. Ε, εντάξει, αυτά δεν παίρνουν τόσο πολλά χρήματα, αλλά αυτό είναι σημαντικό, τα διεθνή δίκτυα. Για το 2012 για το σχετικό προβλογισμό και μετά, εμείς δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από το Συμβούλιο για το τι πρόκειται να γίνει. Υπήρξε κάποια καθυστέρηση, όπως είπατε στην αρχή, από τα κράτη-μέλη για τέτοιου είδους προγράμματα. Γι' αυτό ε, προσπάθησε να γίνει τέτοια μείωση ή απλώς ήταν κάποια ε, φορολογική ανάγκη για να γίνουν αυτές οι μειώσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τελευταίος Γιάνν Όλμπριχτ. Θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό που είπε η κυρία Γένσεν όντω είναι, είναι αλήθεια. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι αντίθετη. Η Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι αντίθετη με ένα ταμείο μεταφορών. Αλλά δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι εμεί θέλουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση και το να μην ε, ολοκληρώνουμε τίποτα είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο ε, δεν γίνεται ή πρέπει να, πρέπει να αποφασίσουμε. Αν δεν θέλουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε οι δικαιούχοι να το κάνουν αυτό σε εθνικό επίπεδο, α γίνει έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το πούμε. Να μιλήσουμε για τη συμπληρωματικότητα των πολιτικών όμω. Γιατί έχετε, έχει οργανωθεί το πράγμα όπω θα έπρεπε. Δηλαδή, το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Επιτρόπος θα, θα σχεδιάσει τη σύμβαση μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών. Και η σύμβαση αυτή θα δια, περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Ο Επίτροπος Μεταφορών θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για να υπάρξει συμπληρωματικότητα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που χρησιμοποίησατε αυτή ακριβώς την έκφραση. Είπατε ότι τα χρήματα δεν είναι στη Ρέτζη, αλλά είναι στα χέρια της διοίκησης και είναι σημαντικό. Είναι διαφορετική όμως αυτή η διοίκηση. Δεν μπορείτε να λέτε ότι τα χρήματα είναι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει επικριθεί πολλές φορές η Επιτροπή αυτή. Οπότε εγώ τονίζω και πάλι τη συμπληρωματικότητα. Ερώτημα, θα υπάρξει κάποια συνέχεια όσον ε, στην ε, όλη διαδικασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ευχαριστώ. Ωραία, οπότε τώρα θα απαντήσει ο επίτροπο. So, I... Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες. Εκτιμώ ιδιαίτερο τη θερμή σας στήριξη προς τον τομέα των μεταφορών. Τώρα, τι μπορώ να πω συγκεκριμένα για τη γενική μας προσέγγιση. Σε αυτήν την περίοδο του έτους είναι η καταλληλότερη στιγμή να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για τα θέματα αυτά οι μεταφορέ μπορούν πραγματικά να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν είναι δική μου εντύπωση. Είναι πολλοί κύκλοι που θεωρούν ε, τις μεταφορές σαν κάτι που ενοχλεί βεβαίω και ω κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όμως τα προβλήματα που προκαλούνται από τις μεταφορές είναι τόσο σημαντικά για όλου, για τόσου πολίτε που δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Μιλάμε για συμφορήσεις, μιλάμε για μετακινήσεις συστηματικές. Το να βελτιώσουμε το κύρος και τη σημασία του τομέα των μεταφορών είναι ένας από τους στόχους μου και θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας και με τα προγραμματικά μας έγγραφα. Αλλά εδώ θα πρέπει να επιδιώξουμε πραγματικά και την αύξηση του βάρους των μεταφορών στον προπολογισμό. Ξέρετε τα θέματα του προπολογισμού πολύ καλά. Κανείς δεν το αρνείται αυτό ότι είναι απαραίτητο. Το πρώτο στο οποίο θέλω να απαντήσω, κυρίως στον κύριο Γέντσεν που το ρώτησε, τι θα γίνει αν δεν καταφέρετε να βρείτε κονδύλια με τα ευρωμόλογα και όλα τα άλλα, εάν δεν γίνει τίποτα. Πολλοί υπεύθυνοι για τα οικονομικά λένε ότι ωραίο είναι να έχει κανείς διαφορετικά προγράμματα, Και βεβαίω, ωραίο θα ήταν να ελπίζουμε ότι τα προγράμματά μα θα μα φέρουν και έσοδα. Όμω το βασικό είναι η, ο προπολογισμό. Η χρήση και εκταμείευση κονδυλίων σήμερα, η χρηματοδότηση των μεταφορών από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Εάν μείνουν τα πράγματα ως έχουν για τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές, για μένα αυτό θα είναι δράμα και θα πλήξει γενικότερα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα ευρωομόλογα στην υπηρεσία μας. Έχουμε προχωρήσει πολύ στις μεταφορές, έχουμε συνεισφέρει όσο περισσότερο μπορούμε στο πρόγραμμα των ευρωμολόγων και έχουμε δώσει πολλές ιδέες για στατικικές κινήσεις, αλλά θα πρέπει αυτό να είναι απλώς ένα συμπλήρωμα. Θεμελιώδεις ανάγκες μας πρέπει ακόμη να χρηματοδοτηθούν και να βρεθούν πηγές χρηματοδότησης. Σας λέμε λοιπόν το εξή: Εάν δεν αυξηθεί συνολικά ο προπολογισμό για τις υποδομές, ας πούμε, όπου λέγεται ότι το μερίδιο των μεταφορών είναι κάτω του 1% για το δικές μας ανάγκες. Αυτό δεν αρκεί προφανώς για, το, για τη διασυνοριακή διάσταση και την προσέγγιση με τα διευρω... για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τα στοιχεία των μεταφορών είναι τα πλέον ζωτική σημασίας. Το βλέπουμε αυτό και στο ισχύον πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Τα διασυνοριακά στοιχεία όλα έχουν καθυστερήσει. Τα εθνικά χρηματοδοτούνται, προγραμματίζονται, τα διασυνοριακά καθυστερούν. Για τα επόμενα διευρωπαϊκά δίκτυα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια σαφή δέσμευση από τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο πολιτικά ανοίγματα, ότι κάποιο θέλει να φτιάξει μια σύραγγα, α πούμε, ένα τούνελ. Όχι. Πρέπει να είναι σαφέ ποιε είναι οι δεσμεύσει των κρατών μελών τι θα χρηματοδοτήσουν. Θέλουμε πίνακες και στοιχεία. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο. Επίσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες είναι ενδιαφέρον ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα έναν κοινό ορισμό. Το πώς θα αποσαφηνίσουμε αυτό το θέμα είναι στα χέρια σας. Το πώς θα, πώς θα συνδυάσουμε τα διαφορετικά ταμεία με τα ταμεία συνοχής στρατηγικά διευρωπαϊκά δίκτυα. Άκουσα εδώ να εκφράζονται αμφιβολίες, ενδιασμοί για τις προϋποθέσεις, τους όρους, για το earmarking. Κάποιοι είναι υπέρ μιας ε, συνεπούς προσέγγισης. Όμως, είναι, κάποια κατημέλη συμμερίζονται σαφέστατα αυτή την άποψη, αλλά κάποιοι είναι καχύποπτοι. Δεν θέλουμε τα κονδύλια της συνοχής ε, να χρηματοδοτηθούν οι περιφερειακοί των πρωτευουσών κυκλικοί. Δεν το θεωρούν πανευρωπαϊκή εμβέλεια πρόγραμμα αυτό. Εμεί στην Επιτροπή και επειδή συνεργάζομαι με τον συνάδελφο Χάν για να βρούμε στις περιφερειακές συμβάσεις εδώ τέτοια στοιχεία, στοιχεία πολιτικής συνοχής, χρειαζόμαστε και τη δική σας τη στήριξη. Αν δεν μας στηρίξετε, δεν θα τα καταφέρουμε. Εάν ναι, κάτι θα γίνει, ίσω όχι κατά 100%, αλλά τουλάχιστον θα αποφύγουμε να λέμε ότι έχουμε πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων, με ό,τι αριθμό, με ό,τι κονδύλι και να έχουμε, και να έρχεται ο υπουργό του κάθε κράτου και να μου λέει, κοιτάξτε, άλλαξε η κυβέρνηση, πάει, άλλαξε, έχουμε άλλε προτεραιότητε τώρα. Χρειαζόμαστε τον τάδε δρόμο στην τάδε περιοχή. Γι' αυτό θα το πάρουμε. Το κονδύλι θα το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε να πάρουμε από τη συνοχή, να πάρουμε από τα διευθυντικά ταμεία για να καλύψουμε τις τοπικές μας ανάγκες. Ε, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι και αστείο και δεν μπορούμε να το αποδεχόμαστε συνεχώς Για τις προποθέσει λοιπόν που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια συνεννόηση κοινή μεταξύ μας αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε και εδώ σε βάθος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος επίση για τις ερωτήσεις που ε, τέθηκαν για τη χρήση των κονδυλίων. Έχω βρεθεί να κάθομαι στην αίθουσα αυτή ως επίτροπος και υπεύθυνο για τις απαλλαγές και για να απαντήσω στις, στην ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών. Είχαμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση των κονδυλίων των διευρωπαϊκών δικτύων. Είχαμε χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ υποθέτοντας ότι δεν θα ε, δαπανηθούν όλα τα κονδύλια. Λοιπόν, νομίζω ότι βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούνται επαρκώς και αποτελεσματικώς τα κονδύλια. Και κάτι που όλοι έθιξαν όσοι παρενέβησαν είναι ότι χρειαζόμαστε και ανάπτυξη των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων και περισσότερη έμφαση στο περιβάλλον. Βοηθήστε μας, βοηθήστε μας να αναπτύξουμε τις σιδηροδρόμους. Χωρίς σιδηροδρόμους δεν θα αλλάξει η χρήση των οδικών δικτύων. Εδώ έχουμε το στοιχείο κλειδί. Χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή πολιτική για τους σιδηροδρόμους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε πολιτικές για την ε, αεροπλοεία, λόγω χάρη. Οι σιδηρόδρομοι πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι άκρος σημαντικό. για την πολιτική συνοχή και τα σιδηροδρομικά δίκτυα και το κατά πόσον καταλήγουμε να συζητάμε το ίδιο θέμα. Ναι, όλοι θα θέλαμε πανευρωπαϊκά προγράμματα, όμως δεν αποκλείουμε το δικό δίκτυο. Ιδίω στα ανατολικά μέρη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το δίκτυο είναι φτωχό. Είναι λοιπές και αυτό έχει και περιβαλλοντικό αντίκτυπο βεβαίως. Λιγότερη συμφόρηση εφόσον υπάρχουν καλά οδικά δίκτυα, άρα και λιγότερη ρήπανση. Δεν μπορεί λοιπόν αυτομάτως να το αποκλείουμε το δικό δίκτυο, όμως σε κάθε περίπτωση θέλουμε να προωθήσουμε μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχουν σαφείς επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές μας βλέψεις και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής μας ε, πολιτικής. Για τον Σέζαρ, ως προς την ανάπτυξη του, και την εκδίπλωση του Σέζαρ, όλα πάνε όπως είχαν σχεδιαστεί. Τώρα, πώς θα υλοποιηθεί ακριβώ το πρόγραμμα αυτό. Αυτό εξαρτάται από τη συνολική ε, μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου της ε, ε, αεροπορικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, χωρίς τέτοια μεταρρύθμιση δεν θα πάνε τα πράγματα όπως είχαμε προβλέψει. Πολλά κρατημέλη όρισαν ε, και προγραμμάτισαν μεταρρύθμιση του δικού τους ε, συστήματος. Μέσα στη φετινή χρονιά ή μέσα και στο πρώτο εξάμεινο της φετινής χρονιάς θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η τάση, αυτά τα σχέδια. Και αν δεν προχωρήσουν σωστά θα δούμε αν πρέπει πραγματικά κάτι να κάνουμε για να έχουμε καλύτερη και, μεγαλ... και πιο ισχυρή διαχείριση της ε, αεροπλοείας για τα καύσιμα. Και αυτό μας απασχολεί. Ελπίζουμε ότι με την καλή μας συνεργασία ή τέλος πάντων με τη συνεργασία με τις Αμερικανικές Αρχές θα καταλήξουμε σε μια κοινή συνεννόηση ώστε να αναπτύξουμε τα κατάλληλα συστήματα και το θέλουμε αυτό γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε αφού έχουν ε, πόρου στρατιωτικού. Αυτό διαφέρει από τι ευρωπαϊκέ μα συνήθειε. Όμω θέλουμε ένα τέτοιο σύστημα που να λειτουργήσει και να μα διευκολύνει, εφόσον βεβαίω προχωρήσουν επιτυχώ οι μεταρρυθμίσει τη ε, διαχείριση τη αεροπορική κυκλοφορία. Το Γαλιλαίο που το έθιξαν ένας-δυο βουλευτές, ε, εκτός από τον εισηγητή, δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας είναι θέμα του ε, Επιτρόπου που είναι υπεύθυνο για τα θέματα βιομηχανία. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω για τα του Γαλιλαίου. Γι' αυτό που ρωτήσατε τώρα, είναι πολιτική απόφαση. Δεν γνωρίζω στον ε, πολιετή μας προγραμματισμό το βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να εξακολουθήσουν έτσι. Χρειάζονται πληρωμές και πιστώσεις να συνδυάζονται. Θα δούμε ποια είναι όλα αυτά τα προγράμματα που θέλουμε να χρηματοδοτηθούν. Όμω θα το ξανασυζητήσουμε άμεσα με τι δημοσιονομικέ αρχέ. Αυτά όλα έχουν να κάνουν και με την αναδιάρθρωση και την αναθεώρηση του που αποδίδονται τα διάφορα κονδύλια. Νομίζω λίγο πολύ. Αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όντως, βεβαίως σήμερα ξαναμάθαμε ότι μπορεί κανείς να έχει καλές ιδέες και όπως μας είπε ο Επίτροπος ε, ε, χρειαζόμαστε χρήματα. Χωρίς τα χρήματα τίποτα δεν γίνεται για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι ιδέες. Γι' αυτό και ε, δεν το αναφέρατε εμένα, αλλά φαντάζομαι ότι μας στηρίζετε όσον αφορά την ιδέα ε, της ε, Προέδρου των, με, της Επιτροπής Μεταφορών ότι ή θα χρησιμοποιήσουμε ή θα χάσουμε τη χρηματοδότηση σχετικά με τα, τις ανατεθειμένες πιστώσεις διότι Εάν δεν υπάρχουν σωστές μεταφορές δεν μπορεί να υπάρχει σωστή εσωτερική αγορά. Οπότε τώρα ο Σαλβαδόρ θα κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ε, ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτή τη συζήτηση που είναι σημαντική και βοηθά τον εισηγητή να καταρτήσει τη θέση του διότι ε, ε, με ενδιαφέρει πολύ τι λέει η αρμόδια επιτροπή ξαναπαίρνω την ξαναχρησιμοποιώ ότι η φράση της Προέδρου δηλαδή αν δεν μπορεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός σας δούμε τι είναι η δομή της κάτω από το 1% του προϋπολογισμού ε, είναι κάτι το οποίο να απευχόμεθα και ε, όσον αφορά τις ε, συγκεκριμένες ε, προτάσεις των συναδέλφων ε, εκτός από το αν μπορεί κανείς να συνδυάσει και να συνδέσει τη Γαλλία με τη Βαρκελόνη υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία θα συμφωνούσαμε δηλαδή καταρχήν ότι χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις που θα διατεθούν στην υποδομή θα έχουν προστιθέμενη αξία και θα τονιστεί ιδιαιτέρως η κάλυψη όλων των διασυνοριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να αποφύγει κανεί την τάση που υπάρχει στα κράτη-μέλη να πρημοδοτούν τις ε, τοπικές υποδομές για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ε, με κάποια συνεκτικότητα τα διευρωπαϊκά δίκτυα με διευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές. Είπατε επίσης ότι ε, τα κράτη χρησιμοποιούν ε, μελέτες για να αξιολογήσουν την σκοπιμότητα των υποδομών τους. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε πόσο, σημαντική μπορεί να, μπορεί, πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο σιδηρόδρομος, διότι υπάρχουν χώρες οποίες υστερούν στις σιδηροδρομικές ε, υποδομές. Πριν ε, λάβουμε λοιπόν ακραίες αποφάσεις ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση χώρα προς χώρα. Χρηματοδότηση που είναι βασική για τις τις μεταφορές και τις σχετικές πολιτικές. Θα πρέπει καταρχήν να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα υποδομών με τα μία συνοχής, με διαρθρωτικά κεφάλαια και σε συντονισμό με την περιφερειακή πολιτική να καταρτήσουμε κοινού στόχους διότι ακόμη αναρωτιόμαστε και δεν νομίζω ότι έχει καθησυχαστεί αυτή η ανησυχία αν δεν θα έπρεπε να έχουμε δεσμεύσει ορισμένα κεφάλαια ή να έχουμε χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικό ταμεία πιο εντατικά ε, σε αυτά τα προγράμματα διότι σας υπενθυμίζω θυμίζω ότι σήμερα το πρωί είδαμε ότι όλοι οι ε, επίτροποι που αναφέρονται σε θέματα δαπανών ε, εύχονται όλες οι πολιτικές να είναι οριζόντιες και όπως και εσείς όπως και ο Επίτροπος ο Χάρμς ζητάμε, ζητάτε να υπάρξουν ορισμένες προποθέσεις θα ρωτήσουμε και τον κύριο Χάρμς στις 10 Φεβρουαρίες, Φεβρουαρίου αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο διότι πρέπει να δούμε αν τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο. Συμφωνούμε με την χρήση των ε, των ε, ε, κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής και τράπεζας επενδύσεως και θα δούμε τι θα γίνει και με τα διάφορα ταμεία αλλά μέχρι στιγμής ε, βλέπουμε ότι όπου υπάρχει συγχρηματοδότηση δεν ήρκεσε η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα εφόσον αυτός βαστίζεται σε άλλα κριτήρια δηλαδή στην ε, κερδοφορία. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο να προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα που είναι προγράμματα υποδομής και καταλήγω με την πολιτική των ε, σιδηροδρόμων διότι ε, σαν εκπρόσωπος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και εμείς ε, προσβλέπουμε ε, σε ε, αηφόρες υποδομές. Άρα χρειάζεται μία πανευρωπαϊκή πολιτική για τους σιδηροδρόμους, διότι μετά από τόσα χρόνια που συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε όντως να υπάρχει. Ενώ ακούμε και μιλούν για το ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο που θα ήταν το αντίστοιχο προς τον ενιαίο αέριο χώρο της Ευρώπης και φαντάζομαι ότι αυτό θα ενισχύσει την ε, ευρωπαϊκή αξία. Γι' αυτό και εσύ, κυρία Πρόεδρε πιστεύω ότι ο ε, Επίτροπος μας ε, πέτρεψε να συμφωνήσουμε σε όλους τους τομείς τους οποίους παρουσιάζεται στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα μπορέσει η Επιτροπή να είναι ένα σύμμαχός μας στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο διότι ε, μπορεί μεταξύ μας να λέμε πολλά αλλά μετά να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ που βρήκατε χρόνο να έρθετε να μας επισκεφθείτε και από κοινού με να συζητήσετε την πολιτική μεταφορών. Κατόπιν αυτού φαντάζομαι ότι μπορούμε ε, να καλωσορίσουμε την επόμενη ε, επίτροπο και ε, θα πάω να την υποδεχθώ στην είσοδο. Όχι συναδελφοί, δεν κάνουμε διάλειμμα. Ποιο σα είπε ότι κάνουμε διάλειμμα. Θα καλωσορίσουμε την Επίτροπο για την έρευνα. Έρευνα, καινοτομία και επιστήμες. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Έχουμε διάφορα ερωτήματα τα οποία τα έχετε δει και γραπτός. Ο εισηγητής μας είναι εδώ και έχει επίσης θέσει και καταγράψει διάφορα ερωτήματα τα οποία θέλουμε να σας απευθύνουμε. Πέντε λεπτά θα πάρει την, ε, το λόγο ο εισηγητής Σας το ξαναλέω, την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Ε, θα λάβετε εσείς μετά το λόγο για 10 λεπτά για να κάνετε μια δήλωση και μετά θα ακούσουμε ένα γύρο παρεμβάσεων από τους προσώπους των πολιτικών ομάδων και ανάλογα με το πόσο χρόνο θα έχουμε θα ακούσουμε και άλλους ομιλητές που, από τους ε, συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις και μετά πάλι θα πάρετε το λόγο εσείς για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ο Σαλβαδόρ έχει και πάλι το λόγο. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ την Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στα τελευταία, στο τελευταίο τμήμα τη πολύ γεμάτη ημερήσια διαταξή μας ακούσαμε τις παρεμβάσεις πολλών επιτρόπων σήμερα για διάφορους τομείς πολιτική που είναι πολύ σημαντικοί όταν πρέπει, εφόσον η δική μα επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την άποψή της για τη δομή και το μέγεθος των ε, επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Ω ε, επίτροπο έρευνα κοινοτομία και Επιστήμης έχετε απαντήσει ε, διάφορα ερωτήματα. Ε, το, το θέμα της ε, προστιθέμενης αξίας στη δική σας, στο δικό σας τομέα είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί μιλούμε για 7% της κοινοτικής, των κοινοτικών δαπανών που πάει στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, το 93% παρέχεται εθνικά. Η σημαντική λοιπόν ερώτηση, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι το σύστημα τώρα είναι καλύτερα από το να έχουμε έναν νέο ενιαίο χώρο ε, έρευνας και ο προϋπολογισμός για των 27 κρατών μελών για την έρευνα θα μπορούσε να ενσωματωθεί στον ευρωπαϊκό και να συντονίζεται όλο αυτό από την Κομισιόν. Στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου είπατε ότι οι δαπάνες για την έρευνα θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον οι ίδιες όπως είναι και σήμερα. Αυτό είναι αρκετά φιλόδοξο σχέδιο δεδομένων και των τάσεων που υπάρχουν ε, και, των αισθη... και της αίσθησης που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα βέβαια μαζί σας, αλλά ε, εσείς πιστεύετε ότι εάν δούμε τα ε, ποσά στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι επαρκή για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην στρατηγική 2020 όταν μιλούμε για την έρευνα και την ανάπτυξη, για την έρευνα και την κοινοτομία ή όχι. Για τις δομές τώρα. Ε, προς το παρόν η έρευνα και η κοινοτομία βρίσκονται στην ίδια κατηγορία δαπανών, αλλά σε διαφορετικούς υπότιτλους. Αυτό έγινε καταρχάς για να είναι πιο εύκολο να δοθούν τα διαρθωτικά κονδύλια ε, στον έναν ή στον άλλο στόχο. Εμείς θα θέλαμε να μας πείτε εάν κατά τη δική σας άποψη και λαμβάνοντας βεβαίως και υπό, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την δική σας ε, ε, εμπειρία, ποιο είναι, ποια είναι η καλύτερη δομή για τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και πώς μπορούμε να συντονίσουμε αυτή την πολιτική με την πολιτική συνοχής, θέτοντας ίσως κάποιο, ένα σύστημα earmarking. Ή θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη συνέργεια μεταξύ της έρευνας και, των, και της καινοτομίας και των σχετικών προγραμμάτων με τα διαρθωτικά ταμεία. Επίσης, όσοι από εμάς ήμασταν στην Επιτροπή Προϋπολογισμού την προηγούμενη θυμία και, ήμασταν, και ασχοληθήκαμε εντατικά με το θέμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, γνωρίζουμε ότι προς το παρόν Υπάρχουν ε, δύο πράγματα που ε, έχουν ξεκινήσει και ένα τρίτο που επίκειται. Πιστεύετε ότι αυτό το Ινστιτούτο Τεχνολογίας έχει την απαραίτητη βαρύτητα ε, για να μπορέσει να επιδράσει αποφασιστικά σε ό,τι αφορά την κοινοτομία στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν επιτυχές. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο όσο πάμε, ό, πλησιάζουμε προ τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα μας πείτε την απόψη σα γι' αυτό. Και επίσης ε, υπάρχει το θέμα της έρευνα και της βελτίωσης ε, της απόδοσης ε, στα προγράμματα τα ερευνητικά. Ε, έχουμε εισηγητή από το Κοινοβούλιο, ο οποίο είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα αυτό και σε σχέση με την ιδέα της απλούστευσης στα πλαίσια του 8ου προγράμματος πλαισίου το οποίο περιλαμβάνεται στην ατζέντα, γιατί ούτω ή άλλω θα εργαστούμε σύντομα και με αυτό. Ε, Επίση, τα προγράμματα, τα ερευνητικά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται ανάλογα με τα αποτελέσματά του ή ανάλογα με τον τομέα τον οποίο ερευνούν. σω η Επίτροπο θα μπορούσε να πει εδώ στην Επιτροπή μα ποιε είναι οι απόψει τη για τα θέματα αυτά, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο σαφή ιδέα για το τι θα πρέπει τελικά, πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι αφορά τη δομή τη ε, έρευνα και των πόρων για την έρευνα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελάχιστοι πόροι για την έρευνα. Τέλεια, τέλεια, Σαλβαδόρ, τέλεια. Πέντε λεπτά. Ε, κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να συζητήσω σήμερα μαζί σας τον καθοριστικό ρόλο που θα έχουν η ε, στρατηγική, ο στρατηγικό σχεδιασμό τη καινοτομίας και τη ε, ε, γνώση στην ε, νέα κοινωνία που θέλουμε να δημιουργήσουμε και από οικονομική άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μιλήσω εδώ για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και για το πώ θα μπορούσε να σχεδιαστεί για να στηρίξει του στόχου μα. Στην ανακοίνωσή τη ε, για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή πρότεινε όλα τα εργαλεία που αφορούν την ανάκαμψη, την έρευνα και την κοινοτομία να συνδυαστούν σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Οι ευρωπαϊκέ δαπάνε για την κοινοτομία και την έρευνα έχουν διπλασιαστεί στο τελευταίο δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετέ, και έω το 2013 θα φτάσει κάνουν θα φτάνει η χρηματοδότηση αυτή στο 7% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα τωρινά και παλαιότερα προγράμματα έχουν ε, βοηθήσει και διευρύνει τις γνώσεις μας για θέματα επιστημονικού χαρακτήρα όπως οι κλιματικές αλλαγές και έχουν ε, βελτιώσει και την ευημερία των πολιτών μας. Λόγω χάρη με την έρευνα θεραπείων για σπάνιες ασθένειες που δεν μπορούν εύκολα να λυθούν σε εθνικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επίσης έχει δώσει τη δυνατότητα για ε, νέα πορίσματα σε καναλωτικές στις περιπτώσεις των καταναλωτών όπως για τα νέα κινητά με τα συστήματα 3G και 2G. Ε, εδώ Έχουμε προβλέψει 10 δις ευρώ για ορισμένα προγράμματα ετησίων, κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 13.000 έως το 2015. Επίσης μπορεί να βελτιώσουμε το διεθνή μας ανταγωνισμό και την δημιουργία εργασίας, θέσεων εργασίας. Οι δαπάνες μας και ο προπολογισμός μας θα έχουν μεγαλύτερο αντίτυπο στην απασχόληση, την κοινωνία απασχόλησης και τον, ε, τη θέση των πολιτών μας σε αυτή την αγορά. Κάθε ευρώ που ξοδεύουμε μετράει. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε καλύτερα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε μεταρρυθμίσεις όπου απαιτούνται. Οι ανταγωνιστές μας όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν στο να αποδεχτούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται στρατηγική προσέγγιση για την κοινοτομία και την έρευνα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Έρευνα και Ανάπτυξη και τα εργαλεία της ε, μπορούν να πετύχουν τους σκοπούς τους. Έχουν την εμβέλεια και το πεδίο που χρειάζεται για να ε, πετύχουν τι κοινωνικέ ανάγκε, την δημιουργία θέσεων απασχόληση, το να γίνουμε διεθνώ ανταγωνιστικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, χρειάζεται το εξή. Ε, να ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να εξυγχρονίσουν, να επικαιροποιήσουν, να ανανεώσουν τα συστήματα ερευνά του. Το ίδιο που να κάνουμε και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά μα συστήματα. Χρειαζόμαστε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό περισσότερη έρευνα και καινοτομία στο κέντρο του προπολογισμού και να υπάρχει μια σαφή απόκριση στου στόχου τη στρατηγική το 2020. Ταυτόχρονα πρέπει πρέπει να ανταποκριθούμε και να καλύψουμε τι ανάγκε μα, τι αδυναμίε μα στο σύστημα δαπανών μα, να γίνουν πιο απλέ, και αποτελεσματικέ ω προ το αντίκτυπο και πιο προσβατέ και διαφανεί. Σύμφωνα με τη δική μα μελέτη και την ενδιάμεση ε, ε, αποτίμηση των ε, προγραμμάτων ΣΥΠ και του 7ου προγράμματο πλαισίου πρέπει να δούμε τα μικρότερα προγράμματα και τα διαφορετικά μέσα δείχνουν ότι δεν έχουμε συνολική στρατηγική. Πρέπει εδώ πραγματικά να πετύχουμε ε, κάποια ορόσημα με τις δράσεις μας. Ε, να είμαστε ριζοσπαστικοί και αυτό να γίνει με την έρευνα και την καινοτομία. Εδώ έχουμε πολλές φορές πολύπλοκες διοικητικέ διαδικασίε, Οι διαφορετικοί κανόνε και διαδικασίε που ισχύουν για τα προγράμματα όλα αυτά αποδυναμώνουν. Δεν επιτρέπουν το συσχετισμό με του στόχου του 2020 και δημιουργούν και δυσκολίε στην κοινωνία. Η έλλειψη ταχύτητα και δυναμισμού για να μεταφραστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα και υπηρεσίε στην αγορά. Η ανεπαρκή διασύνδεση και συμπληρωματικότητα ε, των στρατηγικών μα ε, στόχων με άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία όπω τα διαθετικά ταμεία ή τα εθνικά προγράμματα έρευνα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που να αντιμετωπίσουμε όπω και σαφή αντίκτυπο των αποτελεσμάτων στου πολίτε μα. Όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει σε ένα κοινό στατικικό πλαίσιο να αναπτυχθούν, να συνδυαστούν ε, χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα και την κοινοτομία. Εδώ χρειάζεται μια νέα εμβέλεια και μια νέα όθηση για να αντιμετωπίσουμε τι μεγάλε ανάγκε τη κοινωνία των πολιτών και να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και θέσει εργασία. Εδώ χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο για να στηρίξουμε τι φιλοδοξίε τη Ευρώπη για το 2020 και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, για να ανταποκριθούμε στι ε, νέε αυτέ φιλοδοξίε, θα πρέπει να στηρίξουμε όλη την αλυσίδα τη καινοτομία, από τα εργαστήρια στην αγορά. Αυτό θα μα επιτρέψει να πείσουμε να αποδείξουμε πιστικά μάλλον πώ αντιμετωπίζουμε τι βασικότερε προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μα προσφέρει μια βάση για να πλουστεύσουμε τα προγράμματά μα, κάνοντα τα πιο ελκυστικά για του δικαιούχου και του συμμετέχοντε. Ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την ε, καινοτομία θα μα επιτρέψει απλούστευση εφόσον εργαζόμαστε με ένα σύνολο κανόνων, ε, διαδικασιών και συστημάτων ε, τεχνολογία. Όποιο και αν είναι το χρηματοδοτικό μέσο. Θα έχουμε απλούστευση του πολύπλοκου συνόλου των συστημάτων χρηματοδότηση και του τρόπου να καθορίζουμε το έμεσο κόστο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κατά αποκοπήν ποσά όπου αυτό είναι δυνατόν, αποτελεσ... χρηματοδότηση που να βασίζεται στα αποτελέσματα, ιδίω για τα μικρότερα προγράμματα και η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί πιλωτικά προγράμματα. Όπω όμω ξέρετε, η επιστημονική κοινότητα επικρίνει ιδιαίτερω αυτή την έννοια και την προσέγγιση. Το ε, ε, σημαντικά βελτιωμένο σύστημα επιστροφή των δαπανών επίση πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Πρέπει εδώ να είμαστε προσεκτικοί στο σχεδιασμό, να έχουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα προγράμματα, να ε, ε, μεταλλευτούμε νέε πηγέ χρηματοδότηση που μπορεί να ε, λειτουργήσουν ω μοχλή, όπω οι εταιρικέ σχέσει δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Εδώ τα εγχειρήματα με κοινό κίνδυνο, με κοινή ανάληψη κινδύνου είναι ένα καλό παράδειγμα νομίζω. Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο θα επιτρέψει και την χρήση των διαδοτικών ταμείων ώστε να αναπτύξουμε τη νέα γενιά των υποδομών των ερευνητικών βασιζόμενη στην περιφερειακή εξειδίκευση. Όπω τα γνωρίζετε, έχω δεσμευτεί πλήρω να συμβάλλω στην απλούστευση. Να ε, άρουμε τα περιτά απαγορευτικά που υπάρχουν και να στηρίξουμε τους καλύτερους ερευνητές και επιστήμονες. Εδώ χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων μας και για αυτό το λόγο πέρσι εγκρίναμε μια ανακοίνωση για την απλούστευση της υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό παρουσίαζε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιλογές για να μειωθεί το διοικητικό άχθος για τους δικαιούχους μας. Αυτό το έγγραφο, Πρόεδρε, έχει πυροδοτήσει εντατικότατες διαθεσμικές συζητήσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο με την έκθεση Καρβάλιο που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία πέρσι τον Νοέμβριο συνέβαλε και στήριξε τις περισσότερες από τις επιλογές που παρουσιάζαμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας. Και μας ε, τροφοδότησε και με νέες ιδέες. Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο θα μα επιτρέψει να οδηγηθούμε σε τυποποιημένου κοινού κανόνε σε όλα τα ερευνητικά κέντρα για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να εκμεταλλευτούμε τι βελτιώσει που έχουμε πετύχει ω τώρα, καθώ και να μειώσουμε την πολυπλοκότητα για του ε, συμμετέχοντε και του δικαιούχου. Ένα σύνολο ερωτημάτων βέβαια παραμένουν αναπάντητα, όπω πώ η μελλοντική έρευνα και καινοτομία θα ε, διορθωθεί ω προ του μηχανισμού χρηματοδότηση, ποιε θα είναι οι προτεραιότητε που θα τεθούν και ποια ε, μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να επιδιώξουμε καλύτερα του στόχου τη στρατηγική του 2020 για την κοινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η συμβολή των συμμετεχόντων θα επιδιωχθεί ε, με ένα μεγάλο γύρο διαβουλεύσεων που πρόκειται να διενεργήσει η Επιτροπή. Ε, θα ξεκινήσει όλο αυτό με μια πράσινη βίβλο που θα θέσει τα βασικά ερωτήματα. Η πράσινη αυτή βίβλο πρόκειται να εγκριθεί σύντομα. Ο γύρο διαβουλεύσεων θα κρατήσει έω το Μάιο, όπου θα κλείσουμε μια εκδήλωση στι 10 Ιουνίου και η έγκριση τη νομοθετική πρόταση τη Επιτροπή προγραμματίζεται για το τέλο του 2011. 2011. Εδώ είναι περιττό να επαναλάβω ότι στρεφόμαστε και προ του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων ώστε να μα δώσουν την πολιτική όθηση που χρειαζόμαστε για την καινοτομία. Ε, και αυτό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Πέμπτη. Ε, θα καταλαβαίνετε, κύριοι και κυρίε βουλευτέ, ότι δεν μπορούμε εδώ να παραβλέψουμε και την επερχόμενη τοποθέτηση τη Επιτροπή για το MFF. Γιατί χρειάζεται εδώ μια νέα διάρθρωση, ένα νέο πρόγραμμα για την καινοτομία και την έρευνα, αλλά παρόλα αυτά είμαι στη διάθεσή σα και είμαι πρόθυμο να απαντήσω όλα τα ερωτήματα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν, στι απορίε σα σε αυτή τη φάση τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ξεκινάμε με το γύρο των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Τέσσερα λεπτά έκαστος. Η Μαρία Καρβάγιο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε η πιο πρόσφατη έκθεση ε, δεν ε, παρουσιάζει τους αριθμούς της έρευνας διότι ε, ένα μεγάλο ποσοστό της έρευνας γίνεται εκτός της Ευρώπης και 69% των διπλωμάτων ευρωσπιτεχνίας που ζητούνται προέρχονται εκτός Ευρώπης. Οπότε ο προϋπολογισμός για τα μελλοντικά προγράμματα θα επιτρέψει να ανανεώσουμε το πρόγραμμά μας αυτό πρέπει να αποφασιστεί ε, τώρα και να προχωρήσουμε δυναμικά διαφορετικά το 2020 θα είναι πολύ αργά για να αναστρέψουμε την κατάσταση. Μία ανάταξη ολόκληρου του συστήματος προβλέπει ότι πρέπει να έχουμε καλύτερη ε, συμμετοχή των τριών πλευρών του τριγώνου γνώσεως και να συνδυάσουμε καλύτερα ε, την έρευνα με τους δοσι δημοσιονομικές ε, ε, διατυπώσεις. Θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα. Καταρχάς θα ήθελα να ξέρω πώς, προσπαθεί, προβλέπετε να υλοποιήσετε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ε, τι συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρειαστεί στον τομέα της διασυνοριακής ερευνητικής εργασίας διότι κύριε Επιτροπή Επίτροπε, είχατε αναφερθεί στο έτος 2013. Πώς προβλέπετε ότι θα χρηματοδοτηθούν τα διάφορα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης, ε, ε, τα διάφορα προγράμματα πλαίσιο το CIT και το EIP διότι διαφορετικά δεν βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να προωθήσει αυτούς τους στόχους. Επίσης αναφέρομαι στην απλοποίηση και σε, μάλιστα σε, με δύο πτυχές. Καταρχήν ε, πώς ε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων οργανισμών που ε, διασπέρνουν τους ε, πόρους που διατίθενται στην ε, έρευνα. Θα πρέπει το περίπλοκο αυτό σύστημα να απλοποιηθεί, να υπάρξει ένα πιο απλό σύστημα πλαίσιο το οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εφαρμόζουν. Το δεύτερο μέρος ερωτήσεως μου αναφέρεται στη διαδικασία δημοσιονομικής απλοποίησης ώστε διότι πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα που θα βασίζεται στην απλοποίηση ή στην νομική βεβαιότητα και στην ε, έρευνα και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε ε, να εξασφαλίσετε τους στόχους που έχουμε θέσει στο 8ο πρόγραμμα πλέον. Ja, vielen Dank. Okay. λοιπόν, ο Ιβάιλο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όπως ε, και η συνάδελφός μου κυρία Καρβάλιο είπε πρέπει να επιτύχουμε τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτα πρέπει να αναστρέψουμε την αρνητική τάση για την έρευνα στην Ευρώπη και δεύτερον εσείς πρέπει ε, να ε, μεταφράσετε σε πρακτική τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον τομέα της έρευνας. Και εδώ έχω διάφορα ερωτήματα που έχω να θα για να δω πώς μπορείτε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους διότι μιλήσατε για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο φαίνεται πολύ ωραίο και πολύ φιλόδοξο αλλά θα ήθελα να έχω τη γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο της χρηματοδότησης. Πιστεύετε ότι οι αριθμοί θα είναι δεσμευτικοί, πόσο θα μπορέσουμε ε, να υποκινήσουμε καλύτερα το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ε, να επενδύσουν στην έρευνα. Επίσης ε, πώς μπορεί κανείς να προωθήσει μικρά προγράμματα ή μετριοπαθή προγράμματα. Τι γίνεται με τις ερευνητικές μονάδες, με μικρές εταιρείε που μπορούν να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιστεύετε ότι πρέπει να βασιστούμε στα μεγαλεπίβολα σχέδια ή θα πρέπει να εμπλέξουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά, η απλοποίηση. Εσείς ήδη αναφέρατε την απλοποίηση και θα, εφόσον το συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο και συζητάμε για τις αλλαγές στο δομιοσονομικό κανονισμό, θα ήθελα να γνωρίζω εάν αναφέρεστε όχι μόνο στην ενοποίηση των κανόνων, αλλά σε μείωση του διοικητικού βάρους και ε, ε, ε, τι, τι εννοείται όταν μιλάμε για ερευνητικές δραστηριότητες διότι στον μελλοντικό δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχει έντονη προσπάθεια να μειώσει κανείς τη χρηματοδότησή του και ε, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης σχετικά με την, ε, ε, την διατήρηση της έρευνας στο μέλλον πρέπει να έχουμε τη την ίδια χρηματοδότηση για μεγάλα προγράμματα και για μικρά προγράμματα. Παραδείγματο χάρη τώρα, ε, αν ε, ε, χρηματοδοτήσουμε περισσότερο το ίτερ, αυτό γίνεται εις βάρος άλλων μικρότερων προγραμμάτων. Μήπως θα, πρέπει ε, να έχουμε μια διαφορετική γραμμή για τα πολύ μεγαλεπίβολα προγράμματα και να μην τα να στη, στα εσωτερικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης μήπως ε, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη γραμμή προπολογισμού που αναφέρεται ε, στο πρόγραμμα και την πολιτική του διαστήματος. Ευχαριστώ. Ο Γιάννη για στους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, Επίτροπο. Γνωρίζουμε όλοι ότι η γνώση μπορεί να είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο, το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτουμε στο σκηνικό του διεθνούς ανταγωνισμού. Πιο σημαντικό και από το φθηνό εργατικό δυναμικό οτιδήποτε άλλο προ στιγμή. Αυτό θα πρέπει να αρχίσει να μα ανησυχεί. Διότι σήμερα μόλις ε, είδαμε τους τελευταίους, τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βλέπουμε και για άλλους τομείς. Πριν από δύο εβδομάδες είδαμε μια Ολλανδική εταιρεία που επρόκειτο να αρχίσει παραγωγή οχημάτων ε, που κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα πτώχευσε πριν από κανένα δίμηνο και αγοράστηκε από κινέζικη εταιρεία. Με μια απλή επένδυση ε, ε, εξαγόρασαν οι Κινέζοι έτη επί ετών όπου είχαν επενδύσει οι Ολλανδοί στην έρευνα και την ε, γνώση και την καινοτομία. Είναι σημαντικό λοιπόν η γνώση να μην διαφεύγει στο εξωτερικό, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον πυρήνα τη μελλοντική μα οικονομία θα έπρεπε να βρίσκεται ακριβώ το θέμα αυτό και ταυτόχρονα και στον πυρήνα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι οριζοντίως θα πρέπει σε όλους τους τομείς να συμπεριληφθεί έρευνα και καινοτομία. Όταν δίνουμε στήριγμα στο εισόδημα των γεωργών, να το συνδυάζουμε ακόμα και στη γεωργία με την έρευνα και την κοινοτομία. Και σε άλλους τομείς όπου γίνονται δαπάνες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. Πώς το βλέπετε αυτό που σας λέω. Το πρωί μας είπε ο Πέτροπος Έτιγκερ ότι η έρευνα είναι θέμα του προπολογισμού. Συμφωνώ απολύτως. Εσείς τι γνώμη έχετε. Εάν σκεφτείτε το μέλλον, τα κράτη-μέλη που θέλουν να παγώσουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ποιο θα είναι ο ρόλο του προπολογισμού αυτού στο να έχουμε πολύ περισσότερε δαπάνε για την έρευνα και την ε, ε, ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο ερώτημα, Πρόεδρε η δυνατότητα απορρόφησης που έχουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάληψη των κονδυλίων είναι σοβαρό πρόβλημα κατά την άποψή σας και αυτή τη στιγμή μήπως έχουμε προβολικά πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Και πραγματικά θα, ήμουν ιδιαίτερα, θα ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα να ακούσω τη δική σα την άποψη. Πώ θα γινόταν είχαμε καλύτερη και μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η Χέλγα. Oh. Once again, thank you, dear Commissioner, for your very committed. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τον λόγο σας, για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτό που λέτε. Ε, να έχουμε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Είναι πιο στρατηγικής απόφασης, ε, σημασίας μάλλον απόφαση που έχουμε να λάβουμε. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό διεθνώ από τι ΗΠΑ, από την Κίνα, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Με τι άλλε αναδυόμενε, τόσο μεγάλε ε, και δυνατέ χώρε. Είναι σαφέ αυτό. Ακούσαμε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι όταν τους δίνεται ευκαιρία. Ε. Λοιπόν, εδώ μιλήσαμε για διευκόλυνση της ε, υλοποίησης των εφαρμογών. Να μπορούμε πια να αγγίξουμε όχι μόνο τους ερευνητές αλλά και τους χρήστες, τους πολίτες. Το σκέφτομαι σοβαρά αυτό, γιατί υπάρχουν πολλέ ιδέε για τι εταιρικέ σχέσει ε, ε, στην καινοτομία και την έρευνα. Εδώ χρειάζεται μια νέα θηρίδα. Ε, να μην πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα απλώ, αλλά για μια ξεκάθαρη ιδέα. Να υπάρχει ένα οργανισμό που να τα διοργανώνει όλα αυτά. Οι ερευνητέ να ξέρουν με μεγάλη σαφήνεια και με απλό τρόπο πού θα απευθυνθούν. Να απλουστευτεί η καθημερινή του ζωή. Έπειτα, μια δεύτερη ιδέα για την οποία θα ήθελα κάποια σχόλια, είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εδώ Ξέρετε ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, γιατί το χρειαζόμαστε. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι θα γίνει με την, ε, με την ημερομηνία που θα αρχίσει πλέον να ισχύει αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και ως μέλος της Επιτροπής μας θέλω να τονίσω ότι η δημιουργική βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντική στον τομέα της καινοτομίας των δημιουργικών νέων ιδεών, αλλά, ε, άρα είναι και απόλυτα αλληλένδετες με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έπρεπε να είναι ένα απόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο ερώτημα του κυρίου Γκαρίγκα για τις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας. Και εδώ τι γίνεται. Και μια από τι μεγαλύτερε αντιπαραθέσει μα. Ο κύριο Έτιγκερ το πρωί είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ και της έρευνα. Όμω στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή και με τον προπολογισμό που έχουμε υπάρχει και ε, σύγκρουση και υπάρχει και ανταγωνισμό. Ποια είναι η άποψή σα λοιπόν για αυτό το δυσχερέ και ακαθόδε ερώτημα. Ευχαριστώ. ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καθίσταται σαφές ότι σήμερα τα περισσότερα κονδύλια προκύπτουν από τους εθνικούς κορβανάδες στην έρευνα και την καινοτομία. Όταν θα περάσουμε στο, στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ε, χρηματοδοτεί μεγαλύτερα ποσά από ότι τα κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω ότι τίθεται το ερώτημα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προτεραιοτήτων των κρατών μελών. Σε ποιο βαθμό συντονίζονται αυτές οι προτεραιότητες. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τα κρατημέλη να συνεργαστεί για τον τομέα αυτό έτσι ώστε να επενδύσει σύμφωνα και με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Εσείς πώς το φαντάζεστε, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά που γίνονται στα κρατημέλη με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτά που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μας οι συνδυασμένες πηγές σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η επένδυση σε δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη πρόκληση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν από την ΚΟΕ. Η κυρία Αντρέα όμως είναι εδώ. η κυρία Τζαβέλα θα θέσει το ερώτημα. Thank you, Martha. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, Μάρτα. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει μια ταινία του Hollywood που παίζει στα σινεμά που λέγεται The Social Network η οποία περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο πώς έγινε η τεχνολογική επανάσταση στα πλαίσια της ανάληψης κινδύνου σε καινούριε εταιρείε. Το πιο σημαντικό όμως, στην ταινία αυτή βλέπουμε ότι η επανάσταση του διαδικτύου προέκυψε λόγω του, ότι, λόγω του συστήματος του παγκοσμίου που συνδέθηκε ε, ε, ε, στο διαδικτύο με τα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ένωση Καινοτομίας οι όροι αυτοί, ε, ε, κράτη, ε, καινοτομία, πανεπιστήμια, δεν χρησιμοποιούνται όσο θα έπρεπε. Νομίζω ότι μας λείπει και η κουλτούρα, μας λείπει και η νοοτροπία ενός δικτύου πηγών για την καινοτομία. Το ερώτημά μου λοιπόν μετά από όλα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ε, ε, ε, προγράμματα έρευνας και κοινοτομίας επί τη βάση αποτελεσμάτων παρά επί τη βάση δραστηριοτήτων στη ΣΥΠΑ. Χρησιμοποιούν μεθόδους στατιστικών που καταγράφουν μέσω των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ τεχνολογίας και ε, πανεπιστημίων τα αποτελέσματα ε, αυτών των προγραμμάτων και ελέγχουν τις συνέπειες των επενδύσεων στην ε, καινοτομία, στις, στην υγεία, στην απασχόληση κτλ αυτά τα ε, ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια που δεν έχουν δείξει καθόλου αποτελέσματα παρόλο που έχουν χρηματοδοτηθεί με κρατικά κονδύλια βγαίνουν από τη λίστα και δεν είναι πλέον δικαιούχοι χρηματοδότησης. Ερώτημα μου λοιπόν, γιατί δεν υιοθετούμε και εμείς ένα τέτοιο σύστημα ώστε να έχουμε μία ιδέα, έτσι, μία εικόνα του ποια είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών των κονδυλίων που δαπανούμε για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα ε, ολοκληρώθηκε ο κύκλος ε, των εκπροσώπων των ε, πολιτικών ομάδων. Ε, είτε όλοι όντως πολύ πειθαρχημένοι και τώρα θα ακούσουμε τις πρώτες απαντήσεις από την Επίτροπο. Η Επίτροπος έχει χρόνο μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Θα σας πω ποιος είναι ο επόμενος, ε, η επόμενη. Αγγέλικα Νίμπλερ, Ράιμαρ Μπέγκε, Έκμαν, Πίπερ, Γκοτμάνις και Μέρι Μαγκίνας είναι οι επόμενοι ομιλητές και η Μάρτα Αντρέασεν και ο κύριος Έλλης και η κυρία Γκρέσλε. Ωραία. Αυτή είναι για τον επόμενο γύρο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πρώτο γύρο απαντήσεων από την Επίτροπο. Thank you very much, uh, Chairwoman, and Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όσους ε, πήραν το λόγο και όσους έθεσαν ε, ερωτήματα. Για τα πρώτα, για τα μεγάλα ε, προγράμματα, ITER, Galileo, GMES, όταν εγώ έγινα επίτροπο τον προηγούμενο Φεβρουάριο, είχα να αντιμετωπίσω αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα και περίπλοκο το ITER. Ένα φάκελο που δεν τον είχαμε διαχειριστεί όσο εγώ θα ήθελα, που προέρχομαι και από το ελεκτικό συνέδριο, ένα φάκελο που τα κράτη-μέλη δεν είχαν αναλάβει τίποτα, είπανε πρόβλημά σου είναι κομισιόν το ίτερ και υπήρχαν θέματα διακυβέρνησης, καθώς επίσης και οικονομικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίσαμε το θέμα της διακυβέρνησης, κάναμε αλλαγές στη δομή, στη Βαρκελόνη, ζητήσαμε από τους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν και αυτοί τα θέματα διακυβέρνησή του και την ευθύνη του και να παίξουν το ρόλο που πρέπει. Αλλά η χρηματοδότηση για το ΙΤΕΡ πάντα ήταν το βασικό μας πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι είχαμε βρει μια λύση στον προϋπολογισμό και στις συζητήσεις που έγιναν πριν από τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς ε, υπήρξε ένα πρόβλημα, όπως ξέρετε, με το Κοινοβούλιο, που δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα και αδιέξοδο και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό εμένα μου δίδαξε πολλά. Και είναι κάτι που συνέχεια το προωθώ εντός της Κομισιόν, ότι πρέπει να έχουμε μια, έναν περιορισμένο ε, προϋπολογισμό για μεγάλα προγράμματα υποδομών. Δεν είμαστε καλοί στο να το χειριζόμαστε μόνοι μας, χρειαζόμαστε εμπειρογνωμοσύνη για να γίνει αυτό, αλλά έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη. Κάθε φορά που υπάρχει έλλειμμα στον προπολογισμό, τα κράτη-μέλη στρέφονται στην Κομισιόν. Δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε αυτό να συνεχίζεται. Οπότε εγώ είμαι υπέρ της άποψης που δημιουργήθηκε και λόγω του, του προβληματισμού που προέκυψε με το ΙΤΕΡ, ότι έτσι θα πρέπει να γίνονται από εδώ και μπρος τα πράγματα. Απλούστευση, απλοποίηση. Το επίπεδο χρηματοδότησης ποιο θα πρέπει να είναι. Όπως είπε η κυρία Καρβάλιου, σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις μου έχω μιλήσει για το επίπεδο της χρηματοδότησης για το 2000, ως το 2013. Φυσικά δεν ε, παραβλέπω την υποστήριξη και για μετά το 2013. Αλλά νομίζω ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, όσο μελετούμε τα προγράμματα έρευνας, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε σε όλους, στους πολίτες, στους φορολογούμενους, ότι εμείς δαπανούμε χρήματα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν προστιθέμενη αξία ε, ε, έναντι αυτών που δαπανώνται από τα κράτη-μέλη και ότι δεν συνεχίζουμε τον την, τον πολλαπλασιασμό ε, χρηματοδότησης διαφόρων προγραμμάτων υπάρχουν διάφορα προγράμματα ή τμήματα έρευνα, όπω όπως, ε, ε, το είδα και εγώ όταν προετοίμασα την ακρόασή μου εδώ, ότι το ίδιο πράγμα γίνεται σε 80 διαφορετικά ε, κομμάτια έρευνα, τα οποία όλα χρηματοδοτούνται και κάνουν το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό επίση είμαι ε, τη άποψη ότι πρέπει να ε, συγκεράσουμε, να συντονίσουμε αυτό που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έναν απλό, απλουστευμένο τρόπο και με έναν τρόπο που να δίνει τη νομική ασφάλεια στους εμπλεκόμενους φορείς και στους πελάτες μας. Και νομίζω ότι ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Επίσης, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα ε, του επίγοντος χαρακτήρα της καινοτομίας. Έχουμε μια ευκαιρία τώρα, με αυτή την εβδομάδα, που θα συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το θέμα της καινοτομίας για πρώτη φορά. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία, μέσω αυτών, να ακούσουμε, την, να, να μας δώσουν την ε, στήριξή τους για τον τομέα αυτό, αλλά έχοντας υπόψη και τα εξή. Ένα που το ανέφερε ένα από τους ομιλητές, που είναι η καινοτομία και, ο, και το scoreboard, ο, ο έλεγχος των επιδόσεων για την έρευνα, που δίνει πολλά αριθμητικά στοιχεία για διάφορα κράτη-μέλη, και όσα τα πάνε καλά και όσα δεν τα πάνε καλά, και σε σχέση και με το background αυτού που είπε ο πρόεδρος Ομπάμα την προηγούμενη, την προηγούμενη εβδομάδα στην ομιλία του για την καινοτομία τα αποτελέσματα και η, έρευνα, και η χρηματοδότηση έρευνα βάσει των αποτελεσμάτων. Είναι κάτι που φυσικά θέλουμε να το δούμε πολύ σοβαρά. Αλλά θα έλεγα και το είπα και στην ομιλία μου ότι αυτό είναι κάτι που η ερευνητική κοινότητα και η επιστημονική κοινότητα βάζει ένα τεράστιο ερωτηματικό και ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τίποτα χωρί να του εμπλέξουμε, χωρί να το συζητήσουμε μαζί του και χωρί να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη στήριξή του. Αλλά πρέπει να έχουμε ε, συνείδηση του ότι υπάρχει από την, ε, έχει μπει από την ε, ερευνητική και την επιστημονική κοινότητα ένα, ένα όριο, α πούμε. Είναι λοιπόν μια νοοτροπία αυτή η οποία υπάρχει στο, στη ΣΥΠΑ περισσότερο από, από ότι εδώ. Έχουμε δει πώ μπορεί να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και αυτή είναι πάντα μπροστά και εμεί πάντα προσπαθούμε από πίσω να του φτάσουμε. Είδαμε αυτό το παράδειγμα το οποίο δόθηκε σε σχέση με τι ε, κάτω χώρε. Αυτό συμβαίνει όμω όχι μόνο στι κατοχώρε, αλλά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εταιρείε και στρατηγικέ εγκαταστάσει αγοράζονται από του Κινέζους. Μα πιέζουν, δεν νομίζαμε ότι πριν από 10 ή 5 χρόνια ότι θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια άλματα όπω αυτά που έχουν ήδη κάνει. Αυτό όμω είναι μια πραγματικότητα. Είναι στην πόρτα μα έχουν φτάσει και πρέπει να το δούμε υπάρχουν στρατηγικοί τρόποι τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το μετωπίσουμε όλες αυτές, για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ε, προκλήσεις. Ε, τώρα, σε αφορά την απορρόφηση και τη δυνατότητα απορρόφησης και αν υπάρχει πρόβλημα. Όπως ξέρετε, επιλέγουμε κατά μέσο όρο ένα, με ένα project ανά τρία. Ένα από τα δύο θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ποιότητας. Οπότε, αν έχουμε περισσότερα χρήματα, θα γινόταν να χρηματοδοτήσουμε παραπάνω προγράμματα από αυτά που τώρα λόγω έλλειψη χρημάτων μένουν εκτό. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Εγώ έχω δεσμευτεί έντονα γι' αυτό. Γιατί έχω δει την εξή κατάσταση. Έχουμε μυριάδες, μικρά εργαλεία, προγράμματα κτλ. τα οποία δεν έχουν κανένα συντονισμό μεταξύ τους. Δεν υπάρχει εναρμόνιση των κανόνων, των διαδικασιών. Οπότε, αν εσύ σε μια μικρή εταιρεία, μικρομεσαία, έρχεσαι στην Κομισιόν για να πάρει χρηματοδότηση, θέλει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο, θε να πάρει και χρηματοδότηση από το CIP, ίσω να χρηματοδοτηθεί και από τα διορθωτικά ταμεία κτλ. Πρέπει να πα λοιπόν σε διάφορε θηρίδε για να κάνει την αίτησή σου. Εμεί θέλουμε να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου με συγκεκριμένου κανόνε, οπότε έρχεσαι, αποδεικνύει ότι είσαι μικρομεσαία επιχείρηση, και, και λαμβάνει την επιχορήγηση. Αυτό νομίζω ότι θα είναι μια τεράστια θετική εξέλιξη για την απλούστευση. Δεν είναι αρκετό να λέμε ναι πρέπει να απλουστεύσουμε τα πράγματα και να το συζητάμε θεωρητικά. Πρέπει να αποδείξουμε με τις πράξει μας και με τις προτάσεις μας ότι η απλούστευση θα πραγματοποιηθεί και ότι το διοικητικό άχθος που απομακρύνει όλους από την Κομισιόν τώρα θα μειωθεί δραματικά ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν. Και δεν είναι η Κομισιόν που μιλά για την απλούστευση πολύ καιρό. Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουνα για 10 χρόνια στο ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο σε πολλές φορές σε αιτήσεις εκθέσεις του έχει πει ότι η απλούστευση είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το στρατηγικό πλαίσιο λοιπόν κάνει επίση και κάτι άλλο. Συνδυάζει την, την ερευνητική οικογένεια, αυτό που λέω εγώ. Όταν μιλούμε δηλαδή για ενέργεια, για την ψηφιακή ατζέντα, για την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό, για οτιδήποτε, οποιοδήποτε τομέα είναι αυτός δαπανών για τον οποίο συζητούμε, που περιλαμβάνει έρευνα, χρηματοδότηση έρευνα και στήριξη, όλα θα πρέπει αυτά να αποτελέσουν τμήμα του στρατηγικού ε, πλαισίου. Το EIT είναι ένα παράδειγμα φορέα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμβολή 300 εκατομμυρίων ευρώ υποτίθεται ότι θα υποστήριζε την καινοτομία και την έρευνα και την εκπαίδευση και σχετικά προγράμματα και δόθηκε, ε, του δόθηκε μια, ένας βαθμός ανεξαρτησίας, δεν είναι δική μας δηλαδή ε, ε αρμοδιότητα το φορέας αυτό είναι της Επιτρόπου Βασιλείου, αλλά μπαίνοντα στο ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο, έχει το δυναμικό να αναπτυχθεί και να κάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Οπότε δεν είναι απλώς ένα ορφανό παιδάκι στην άκρη, όπως συχνά το, το λέω, είναι κομμάτι του στρατηγικού πλαισίου και επιτρέπεται, μπορεί να, να συνεχίσει με το δικό του ανεξάρτητο αυτόνομο τρόπο τις δραστηριότητε του. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αναπτυχθεί με συνεκτικό και πλήρη τρόπο, ο οποίος αποφασίστηκε από την αρχή και ο οποίος ε, κατατέθηκε από την αρχή. Για παράδειγμα, αν δούμε την, ε, το Energy Kick, είναι το μόνο, ε, η μόνη ενιαία φθυρίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με το θέμα της βιώσιμης, ανάπτυξης, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, έχει τα, την απαραίτητη κριτική μάζα για την οποία συζητήσαμε για να λάβει υπόψη όλες, όλη την αλυσίδα από, ε, για την ενέργεια από την παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση μέχρι την διανομή και το λιανεμπόριο. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού που θέλουμε τελικά να κάνουμε με την έρευνα και την καινοτομία στην Κομισιόν. Σε σχέση τώρα με τα διαρθρωτικά ταμεία, νομίζω ότι υπάρχουν συνέργειες στην χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, καινοτομία και ε, έρευνα και των διαρθρωτικών ταμείων. Ξέρω ότι ο Επίτροπο Χαν είναι πολύ, ε, το έχει, πάρει πάρα πολύ σοβαρά το να εξασφαλίσει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί αυτό που εγώ ο, ονομάζω μια σκάλα προ το μια κλίμακα αριστεία. Ε, νομίζω ότι ε, πολλές φορές ακούμε να αναφέρονται προκλήσεις στον τομέα της αριστείας και της ε, έρευνας. Θέλουμε να έχουμε άριστους ερευνητές, θέλουμε να έχουμε άριστους επιστήμονες, αλλά δεν θα διατηρηθούν, δεν θα μείνουν στα κρατημέλη εκτός αν τους δοθεί η άριστη υποδομή που θα τους βοηθήσει να κάνουν τη δουλειά τους στα κράτη-μέλη. Οπότε πρέπει και εμεί να βρούμε τον τρόπο να ενισχύσουμε, να υποστηρίξουμε αυτού του ανθρώπου. Πρέπει να είμαστε σε θέση πάντα να υποστηρίζουμε την αριστεία. Κάνοντα αυτό, πρέπει να βρούμε και τρόπο να βελτιώσουμε την αριστεία, να την ε, διευρύνουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο Ευρωπαϊκός Χώρος έρευνα είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά των όσων είπανε τα μέλη σα. Ε, πολλαπλασιασμό. Ε, δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή σε, στα αυτά που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτά που γίνονται σε εθνικό επίπεδο και είπα και πριν ότι δεν θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε αυτό που καλύτερα γίνεται σε εθνικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε οτιδήποτε κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αντίθεση με αυτά που γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Να μην χρηματοδοτούμε απλώς για να χρηματοδοτούμε, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει προστιθέμενη αξία την οποία ζητούν και οι πολίτε μας. Ίσως, Πρόεδρε, να πρέπει να σταματήσω εδώ για να ακούσουμε και τι υπόλοιπε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντως βλέπουμε ότι είσαστε πολύ ενθουσιώδης, έχετε μία σταθερή πορεία και πρέπει να σας πω ότι μπορούμε ε, έτσι να ε, ε, υποφεληθούμε της παρουσίας σας διότι ε, όταν ε, χρειαστεί να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και να τσακωθούμε για τον προϋπολογισμό μας, για το μελλοντικό προϋπολογισμό, ε, χαιρόμαστε διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται στο πλευρό μας ε, απέναντι στο Συμβούλιο. Τώρα το λόγο έχει η Αγγέλη Νίμπλερ για δύο λεφτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχήν σας ευχαριστώ Χαίρομαι γιατί είπατε και πάλι ότι τα μεγάλα προγράμματα Ήτερ, Γαλιλαίο ε, βρίσκονται σε μία σταθερή βάση και φαντάζομαι ότι έχετε όλη τη στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως για την απλοποίηση. Ε, δηλαδή να έχετε μία πύλη εισόδου για όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας παραδείγματος χάρη. Επίσης είπατε ότι η ανάλυση απέδειξε ότι ε, πολλά μικρά προγράμματα δεν ε, στηρίζονται πολύ αποτελεσματικά. Η δικιά μου παράκληση είναι στο μέλλον να μην προωθούμε μόνο τα μεγάλα προγράμματα στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει και από μικρά προγράμματα τα οποία πρέπει να στηρίξουμε και γι' αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας. Πρέπει και τα πανεπιστήμια και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να υποφεληθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και σχεδόν τελειώνω. Είπατε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων των ερευνητικών με τα ευρωπαϊκά. Φαντάζομαι ότι πολλά έχουν αναδιαταχθεί και ξεκινήσει. Υπήρχε ένα joint programming το οποίο είχαμε επινοήσει για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για να, ε, ε, ε, για να συνδυάσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα με τις εθνικές γραμμές χρηματοδότησης. Έχετε κάτι να μας πείτε σχετικά με αυτό το θέμα και πώς θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε και να μην στηρίζει κανείς σε εθνικό επίπεδο μόνο ό,τι αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Ευχαριστώ αυτό την Επίτροπο γιατί έχουμε μία πολιτική επιμορφωτική η οποία μας επιτρέπει να συνεργαστούμε και διαπιστώνω ότι η πολιτική καινοτομία δεν είναι μόνο μία προέκταση της έρευνας αλλά μία δυνατότητα χρησιμοποιήσεως των δημοσιονομικών πόρων ακόμη και αν τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν τόσο καλά. Θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία αλλά συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι ένα μέρος της καινοτομίας βασίζεται στην πρακτική και πολλές φορές μπορεί να προκληθεί από τους πελάτες μας οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους πόρους Ήδη έχουν διατυπωθεί διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική συνοχή, την οποία θεωρούμε σημαντική. Και δεν μπορεί η πολιτική συνοχής να προωθηθεί στην Ευρώπη χωρίς καλή, καλό συντονισμό. Θα πρέπει πέραν της πολιτικής συνοχής να προωθήσουμε τις περιφέρειες και τα κέντρα γνώσεων. Και τέλος θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας. Πρώτον, πώς μπορούμε να ε, να διαφοροποιηθούμε από τους πόρους των ε, περιφερειών. Πώς μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα που να είναι ενδιαφέρον και πέραν της Ευρώπης. Πώς μπορούμε επιπλέον ε, να ε, ε, επινοήσουμε ε, έξυπνα προϊόντα. Εδώ δηλαδή αναφέρομαι στην καινοτομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και πόσο μπορούμε να συναντηθούμε καλύτερα όσον αφορά τα προγράμματα. Αν συζητάμε για περιφερειακά προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με ερευνητικά προγράμματα. Εδώ υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά, αλλά θα ήθελα να μου πει η Επίτροπος πώς αντιλαμβάνεται την ε, καινοτομία επί της βάσης των πρακτικών εφαρμογών. Ωραία ημερινό ο επόμενος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για τις ε, ενθαρρυντικές απαντήσεις. Συμφωνώ με αυτά που είπαν συνάδελφοι για την ε, χρηματοδότηση των μεγάλων προγραμμάτων τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε και για την ε, προγραμματική περίοδο και θα πρέπει να γνωρίζουμε σαφώς πώς μπορούμε να τα ανεξαρτητοποιήσουμε από τους ετησίους προϋπολογισμούς. Και μετά το ΙΤΑΡ και το τον υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο συνεπάγεται αυτήν την χρηματοδότηση γιατί η έκθεση Καρβάλιο είναι μια πολύ καλή ε, δυνατότητα απλοποίησεως διότι βλέπετε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε εάν προχωρήσουμε ε, από κοινού αλλά έχουμε τα αποτελέσματα του ελεγκτικού συνεδρίου για την έρευνα Εάν λοιπόν ζητήσουμε περισσότερους πόρους για όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της ερεύνης θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση για μία πράσινη κάρτα παρόλο που θα ζητήσουμε περισσότερους πόρους και όλοι έχουμε συμφωνήσει για το κατόφλι το 3%. Ε, ε, σχετικά με το 3% και θέλω εδώ να συγχαρώ τη γραμματεία για το έγγραφο εργασίας το οποίο μας έδωσε και βλέπουμε ότι ε, βρισκόμαστε κάτω από το 2% δηλαδή μας λείπει 1% στην Ευρώπη. Τι θα γίνει με αυτό επίσης πλέον του εβδόμου προγράμματος πλαισίου μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μία ανάλυση και να δούμε πόσο μεταξύ επικουρικότητος και προστιθέμενης αξίας να συντονίσουμε τις εθνικές προσπάθειες ε, να προσθεθεί το ευρωπαϊκός χώρος όπως τον αναφέρατε και επιπλέον όπως είπατε και εσείς η φορολογία πολιτική και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω βάσει της πείρας που έχετε για τα συγκεκριμένα προγράμματα τι από αυτά υπάγονται ή στο μέλλον και πού χρειάζεται να καταρτήσουμε νέες προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Η Λένα Έκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ως συντονίστρια της ΙΤΡΕ έχω ορισμένες παρατηρήσεις και σχόλια και μερικά σύντομα ερωτήματα στο τέλος. Πρώτα απ' όλα βρίσκω ότι υπάρχει ελάχιστο συντονισμό μεταξύ τη στρατηγική για το 2020 και του προγράμματο πλαισίου. Καθώ και άλλων προγραμμάτων με πολιτικέ προθέσει, όπω αναφέραμε. Επιπλέον, δεν ξέρω για τους ελέγχους αν πρέπει να βασιστούμε μόνο στην εμπιστοσύνη, αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε πρακτικά αποτελέσματα, γι' αυτό να μας καθοδηγήσει. Για την απλούστευση, ορισμένα από τα προγράμματα, για ορισμένα από τα προγράμματα έχουμε βασιστεί στους υπάρχοντες κανονισμούς και βλέπουμε πώς μπορούν κάποιοι να χρησιμοποιούν την φαντασία, την εξυπνάδα τους και την ευφύεια τους για να βρίσκουν μέσα εκεί που ο κανονισμός δεν δίνει ευκαιρίες. Ε, εδώ λοιπόν στηρίζω πλήρως την ιδέα σας για το στρατηγικό πλαίσιο, όμως δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνον στον ισχύοντα κανονισμό της Επιτροπής. Δεν θα φτάσει, θα είναι υπερβολικό κάτι τέτοιο. Ε, οργανώσαμε μια ακρόαση στην Ήτρε για την απλούστευση. Και θα πρέπει να δούμε το εξή. Όταν κοιτάζει κανεί αυτά τα στατιστικά δεδομένα και συγκρίνει Ευρώπη και Ηνωμένε Πολιτείε μόνο για τι δημόσιε δαπάνε, εάν προσθέσει και τι ιδιωτικέ και δείτε τη διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπη, είναι τεράστια η απόσταση. Αγεφύρωτο το χάσμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε εάν μπορούμε να στηρίξουμε τις επενδύσει επενδύσεις, επιχειρήσει που να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα που είχαμε μόνο κατά 18% τα τελευταία χρόνια. Το αντίθετο θέλουμε. Άρα η απλούστευση θα πρέπει να απασχολήσει και τη δική σας επιτροπή, την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Πρέπει να είναι άκρα σημασία και για εσά. Για το ΙΤΕΡ. Το θέμα με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι το καθορίζει, το διέπει η συνθήκη Ευρατόμ. Ενώ εμεί ε, πρέπει να προβλέψουμε τα κονδύλια. Αυτοί που αποφασίζουν να βρουν τα χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να πρικοδοτηθεί το ΙΤΕΡ για να δώσει τα αποτελέσματα, να προχωρήσει. Και να μην έχουμε και υπερβολικέ δαπάνε όπω την τελευταία φορά. Και επίση, ποια είναι η άποψή σα για την ενημέρωση. Είναι δυνατόν να έχουμε ενημέρωση στου ιστοτόπου για το πώ προχωρούμε, τι γίνεται, τι πρόοδο έχουμε στην έρευνα. Τέλο, συμφωνώ απολύτω με τι απόψει σα για το EIT. Ε, προχωρεί, λειτουργεί, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά θα τα λύσουμε. Ευχαριστώ. Nächstes Markus Pieper, bitte. Ja, danke. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τις πολύ καλές παρατηρήσεις. Δύο ερωτήματα έχω. Ένα για την ενισχυμένη διασύνδεση διαρθρωτικής πολιτικής και πολιτικής έρευνας. Στις περιφέρειες βλέπουμε πολλά παραδείγματα με την ευρωπαϊκή αριστεία της έρευνας στα γυμνάσια να συμβαίνουν διάφορα και πριν ακριβώς το, το Πανεπιστήμιο να δημιουργούνται διάφορα ερευνητικά κέντρα, τα οποία ακριβώς για το ίδιο θέμα παίρνουν διαρθρωτική ε, χρηματοδότηση. Η κοινοτομία λοιπόν και η έρευνα ε, ε μετακυλίεται στις ε, περιφέρειες μέσω των χρηματοδοτήσεων από το διευθυντικά ταμεία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το σύστημα αυτό και ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και τον μοχλό πίεση για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και ίσως θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Τα διευθυντικά ταμεία ως μοχλό για την ευρωπαϊκή έρευνα. Πολύ πιο έντονα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και ένα ερώτημα πώς, ένας, πώς θα είναι ένα σύστημα, πώς θα έχει όπου θα πρέπει να συνδυάσει αντί, αντίθετες ε, προσδοκίες, πώς θα μπορέσει να συγκεράσει ε, τομείς οι οποίοι τίθενται ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεύτερο ερώτημα. Μιλήσατε για την απλούστευση. Πολλά προγράμματα υπάρχουν και είπατε ότι θέλετε να υπάρχει μόνο μία θηρίδα όπου θα μπορεί ο ετών να λαμβάνει τις ε, πληροφορίες του. Ωραία, η ιδέα καλή είναι. Αλλά πού θα είναι αυτή η θηρίδα, στις Βρυξέλλες, στην περιφέρεια, και ποιο θα είναι αυτό που θα εξυπηρετεί, ποιο θα λαμβάνει την απόφαση πίσω από τη θηρίδα. Πώ ακριβώ, συγκεκριμένα το φαντάζεστε. Ευχαριστώ. Εγώ. Κύριε Πόλσεν, ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που είναι εδώ η Επίτροπος. Θέλω κι εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα που ίσως να μην αφορούν κατά ανάγκη την Επίτροπο, αλλά είναι θέματα που πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Αν, θέλουμε, ε, αν δούμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και αν δούμε και τις ε, τεράστιες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κλιματολογικές αλλαγές, η Ευρώπη εκεί έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και θα συνεχίσει να το έχει και στο μέλλον όταν ε, αντιμετωπίζουμε θέματα κλιματολογικά γιατί είμαστε ένας από τους χώρους που μπορεί να παράγει ε, τρόφιμα. Είμαστε καλή παραγωγή λοιπόν ε, τροφίμων. Υπάρχουν βεβαίως ε, πολλά προβλήματα στα οποία θα έπρεπε να, επι, να, επι, να στοχοθετούμε την έρευνά μας. Ας πούμε, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων διοξιδίου του άνθρακα ε, να έχουμε μια ε, οικονομία χαμηλού άνθρακα, να υπάρχει αντιστάθμιση με οικονομικό για κάθε ε, κιλό τροφίμου που παράγεται, να υπάρχουν δίκαιες πληρωμές για τους γεωργούς, αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων επίσης. Πρέπει να υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικά σημαντικές δυνατότητες ε, χρήσης ε, ζυζανιοκτώνων για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα στο γεωργικό τομέα. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστούμε και θα πρέπει να αφιερώσουμε και χρόνο και χρήμα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε ε, μελλοντικέ ελλείψεις τροφίμων θα πρέπει σήμερα, αύριο, μεθαύριο να αρχίσουμε να μιλούμε για το θέμα των τιμών. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την βιοτεχνολογική έρευνα γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε την ε, βιοτεχνολογία στη Μονσάντο. Έξι μεγάλε εταιρείε είναι υπεύθυνε για, ε, για το 90% τη έρευνα στη βιοτεχνολογία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μεγάλε επενδύσει σε ε, ανεξάρτητου ερευνητέ οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν τι λύσει για τι οδιέ τι οποίε χρειάζονται οι πολίτε όχι απλώς ε, να παραγωγή εισοδιών η οποία δίνει μεγάλο ε, κέρδος. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοθεί όλο αυτό, αν μπορεί να πάει στον ε, ε, προπολογισμό για την ε, γεωργία ή στον προπολογισμό για την έρευνα, πού, πού ανήκει. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η πρακτική κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήβας Κουμάντνης. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα, κυρία Επιτροπέ, που με ανησυχούν λίγο. Όταν δούμε το έγγραφο στη σελίδα 6, λέει ότι η δημόσια χρηματοδότηση είναι 96,2 δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Πολύ περισσότερο από την Κίνα, την Ιαπωνία ή άλλε χώρε. Εκεί είναι πολύ, πολύ χαμηλότερη η χρηματοδότηση. Ερώτημα. χαμηλοτερη χρηματοδοτηση εμεί από, δημόσια, από το δημόσιο κορβανά δίνουμε περισσότερα από, την, ε, από τη ΣΥΠΑ, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και σωστά αποτελέσματα. Ε, ε, αλλά ακούω ότι δεν έχουμε καλά αποτελέσματα, οπότε πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Επίσης, μίλησα, η κυρία Εκ μίλησε για το θέμα της ε, ιδιωτικής ε, επένδυσης. Υπάρχουν μεγάλες ε, συνέπειες μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων γιατί δίδονται τελείως διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία, ειδικά από τα νέα κράτη-μέλη. Ίσως να πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για αυτό. Η ιδιωτική χρηματοδότηση, ας πούμε, για την έρευνα και την ανάπτυξη δεν είναι τεράστια από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, διαφέρει. Επίσης, είδα την παρουσίαση πέρσι τον Νοέμβρη όπου ο βαθμό επιτυχία για τους ε, επιστήμονες ήταν, για την επιστήμη μάλλον ήταν 21%. Είναι τελείω διαφορετικό αυτό από, την, από τα διευθυντικά ταμεία του Ταμείου Γεωργία. Γιατί δεν μιλούμε για earmarking εδώ. Δεν υπάρχει αποθεματικό για τα κράτη-μέλη και για του επιστήμονέ του. Ξεκινώντα όμω από το 2000, αυτό είναι μοναδικό, είναι πρωτοφανέ. Ένα επιστήμονα μαζί με έναν άλλον μπορούσε να κάνει ένα κονσόρτσιο α πούμε. Από το 2007 μέχρι το 2010 ε, πήγανε 275.000, ε, υπήρξαν 275.000 συμμετοχές ε, ε, επιστημόνων. Και το εκπληκτικό ήταν ότι δεν έχει σημασία ποιο ήταν το τμήμα του ΑΕΠ ε, σε εθνικό επίπεδο. Δεν συνδυάστηκε καθόλου αυτό με τον βαθμό επιτυχίας. Δηλαδή, αν, δίνουμε λιγότερα, αλλά βρούμε καλά κονσόρτσια έχουμε πάλι τον ίδιο βαθμό ε, επιτυχίας με, τα, με, την, με το όταν ε, ε επενδύαμε σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης, οι διαρθωτικά ταμεία και επικαλύψεις με, τη, με το πρόγραμμα πλαίσιο και τα προγράμματα έρευνα. Κάποιοι επιστήμονε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα διορθωτικά ταμεία γιατί είναι πιο εύκολο να πάρει κανεί χρήματα από εκεί από άλλα προγράμματα. Και ειδικά σε προγράμματα που κρίνονται από επιστήμονε και όχι από γραφειοκράτε. Είπατε ότι θέλετε να φτιάξετε μια κλίμακα προ την αριστεία, αλλά πώ ακριβώ θα γίνει αυτό δεν είναι απόλυτα σαφέ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα την αρχή της παρουσίασής σας. Απλώς ορισμένα σχόλια. Ίσως όλοι εδώ στην αίθουσα να κατανοούν τα προγράμματα πλαίσιο και πώς λειτουργούν. Εγώ προσπάθησα να το μάθω γιατί βρίσκω το χώρο πολύ περιπλοκό και αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να αλλάξουμε κάποιους όρους. Απλούστευση ας πούμε. Και στη Γεωργία το συζητάμε και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, να σπάσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία και να την παρακολουθήσουμε. Το θέμα είναι υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη σε διάφορετικούς τομείς θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Νομίζω ότι σε κάποια κατημέλη ισχύει αυτό, σίγουρα όχι σε όλα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξέρουμε ότι τα χρήματά μας έτσι δεν ταπανώνται για περίπτωση σκοπού. Επίση, ε, στηρίζω τι προσπάθειέ σα να έχουμε επιστήμονε σε όλη την Ευρώπη που να διασυνδέονται καλύτερα. Αυτό όλο και πιο πολύ το προσεγγίζουμε, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετέ οι επιστημονικέ διασυνδέσει. Επίση, η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξή. Η διασύνδεση με τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, νομίζω. Όλε οι αναπτυγμένε χώρε έχουν αποτύχει στην γεωργική έρευνα και τη μεταφορά γνώσεων. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα έχουμε μια σοβαρότατη αποτυχία. Ήθελα λοιπόν τι απόψει σα και πώ αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και εκτό και παρόλο που ένα συνάδελφο που έκανε αυτό το σχόλιο έφυγε από την αίθουσα, ενώ το είχε θίξει αυτό, η διασύνδεση τη χειροτομία με τις επιδοτήσει του γεωργού. Εδώ μιλάμε για το 50% των επιδοτήσεων σε σχέση με του υπόλοιπου τομεί. Μην θεωρούμε τον, ε, τον προπολογισμό τη Γεωργία ως ένα εύκολο στόχο. Δεν μπορεί εκεί να ξεσορροπήσουμε τόσο δεν κάνουν πολιτικέ. Στο παρελθόν κάναμε πολλά σφάλματα εκεί. Να προσέξουμε μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον και πολλοί θα διαφωνήσουν με αυτό. Και πέραν τη γεωργία. Νομίζω για τη βασική έρευνα έχουμε όλη αυτή την ε, οικολογική οικονομία που ξέρω ότι την ε, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί χρειάζεται λοιπόν να προσεγγίσουμε κι άλλου ε, για να υπάρξει πρόοδο. Η κυρία Αντρίασεν, χωρίς μικρόφωνο. Πριν από 7 χρόνια, όταν αυτό το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμαζαν το πολιετές ε, πρόγραμμα πλαίσιο πολλές ε, ανησυχίες είχαν εκφραστεί που παραμένουν οι ίδιες με αυτές που είχαμε εδώ χρησιμοποιώντας και τους ίδιους όρους στρατηγική ανάπτυξη εργασία, θέσεις εργασίας απλοποίηση και προστιθέμενη αξία δεν έχουμε σαφείς ε, δείκτες για το πόσο αποτελεσματικό υπήρχε αυτό το πρόγραμμα αλλά σήμερα δεν έχουμε ούτε ανάπτυξη ούτε θέσεις εργασίας ε, και ε, πολύ υψηλές τιμές έχουμε τις ετήσιες εκθέσεις το ξέρετε και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές παρατυπίες. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο ε, ότι τα προγράμματα δεν υπήρξαν τόσο επιτυχή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι διαφορετικό. Τι θα αλλάξει αυτή τη φορά. Επίσης ε, διατυπώνται προτάσεις για το 2014 αλλά έχουμε ακόμη τρία χρόνια και υπάρχει και η κρίση σήμερα και η ανεργία που υπάρχει σήμερα. Τι θα γίνει λοιπόν, ε, τι θα συμβεί σε αυτά τα τρία επόμενα έτη ή θα περιμένουμε απλώς μέχρι το 2014 για να βρεθεί η λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τις πολιτικές των διαφόρων κρατών μελών χωρίς να προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε τόσο πολύ εφόσον δεν έχουμε όλους τους πόρους τους οποίους χρειαζόμαστε ο καθορισμός του ποσοστού συντονισμού και ε, κεντρικής συγκεντρώσεως είναι κλειδί ε, για μία τέτοια ε, προσαρμογή στην εποχή της οικονομικής κρίσεως. Ευχαριστώ. Ο James Ellis τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω τρία σημεία τα οποία επαναλαμβάνουν αυτά που έχουν πει οι προλαλήσαντες αλλά με διαφορετικό τρόπο. Μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τη συζητήσαμε σήμερα και στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε ε, ε, να παρουσιάσετε πριν ε, βάλουν αριθμούς στις προοπτικές στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, στη, ε, στον απολογισμό των προγραμμάτων σας για να ξέρετε εάν ε, έχει υπάρξει επιτυχής η η πολιτική που έχει εφαρμοστεί αντί να χρηματοδοτήσουμε αποτυχίες και να διδαχθούμε από, τις, από τα προβλήματα του παρελθόντος. Επίσης 13.000 ερευνητές από τις 200.000 ερευνητών λέγουν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο ε, ε, έρευνας λόγω των συνθήκων υπό τις οποίες εργάζονται. Έχω έναν δικό μου ψηφοφόρο ότι μία ένας ένας ερευνητής χρηματοδοτήθηκε και τώρα του ζητούν να δώσει πίσω τα χρήματα. Άρα υπάρχει πρόβλημα όπως είπε ο Ράιμερ και ε, πώς θα μπορέσει να είναι επιτυχής μία προσπάθεια όταν δεν ξέρετε πώς θα σας δώσουν για να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά σας. Ε, η απλοποίηση. Μήπως ε, οι χώρες δεν θέλουν να χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτυχθούν.

Ε, όσον αφορά το έγγραφο το οποίο δόθηκε πριν από 10 δευτερόλεπτα λέγεται ότι η χρηματοδότηση ε, του Ταμείου Συνοχής επιζητεί την αριστεία χωρίς ε, να επιζητεί την συνοχή που θα έχει και προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι για να είμαστε ειλικριτείς πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε και με ποιον. Διότι είπαμε ότι υπάρχουν ε, υπόλοιπα στον προϋπολογισμό ε, έρευνας διότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Οπότε ε, θα πρέπει καταρχήν να σημειώσουμε την αλλαγή στο ε, ε, εσωτερικό κανονισμό του προσωπικού. Αυτό είναι μία πρώτη αλλαγή. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, νέα πρότυπα τα οποία εφαρμόζουμε, τα οποία δεν μας ικανοποιούν. Ζητούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τράπεζες, τρίτους χρηματοδότες, και μπορώ να σας πω από την Επιτροπή Ήτρε όπως το είπα και εκεί ότι δεν πρόκειται να έχουμε καλά αποτελέσματα διότι δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Άρα τι προσωπικό χρειάζεται ε, βάσει της ε, χρηματοδοτήσεως την οποία μας αναφέρατε σήμερα. Ευχαριστώ η Τερέζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά όσα υπόθηκαν ως τώρα. Και εγώ θα είχα να πω περίπου τα ίδια πράγματα. Με συγχωρείτε αν καθυστέρησα κάπως. Ήμουν όμως και σε μια άλλη επιτροπή. Και έπρεπε να συμμετάσχω και εκεί. Γνωρίζετε ότι ασχολούμαστε με μια σειρά ζητημάτων που καλύπτουν από την έρευνα μέχρι την εκπαίδευση και την κατάρτιση και την γνώση και καινοτομία. Δεν άκουσα όμως να γίνεται λόγος για τους ανθρώπινους πόρους. Σε τι χρησιμεύει να διεγκώσουμε τον προπολογισμό αν δεν έχουμε επιστήμονες και ερευνητέ. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο διαπιστώσαμε ότι λείπουν 700.000 νέοι ερευνητέ αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε επιτελέσει πρόοδο, αλλά όχι αρκετά. Ούτε στην κινητικότητα, ούτε στην ενιαία σταδιοδρομία των ερευνητών. Το θέμα είναι εάν θα πείσουμε τους νέους να επιλέξουν επιστημονικές σταδιοδρομίες. Το πρόγραμμα που σχολιάσατε ε, και αυτό που ανέλαβε η συνάδελφος που ήταν επιφορτισμένο και με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Μίλησε για κέντρα αριστείας, αυτό έδωσε κάποια αποτελέσματα και ακόμη λειτουργεί. Αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερος. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να κατανείμουμε πιο ισότομα, ισότιμα τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες. Να μην υπάρχουν διαχωριστικά βορρά και νότου, ανδρών και γυναικών, φτωχών και περισσότερων χωρών. Εδώ λοιπόν, αν θέλουμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη βοήθεια, στη βοήθεια των χωρών που ακόμη ε, βρίσκονται σε καθυστέρηση. Και τώρα φτάνω στο ερώτημά μου. Πότε θα επιλύσουμε το θέμα της έλλειψης επιστημόνων και ερευνητών στην Ευρώπη και τι θα κάνουμε χωρίς να μας ε, διαφύγει τίποτα από την αριστεία που τόσο χρειαζόμαστε και τέλος υπάρχουν δύο μέσα, δύο προγράμματα που έχουν θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσουν για το μέλλον. Και την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Το ένα είναι το πρόγραμμα η IT και το άλλο είναι το ΚΙΚ. Οι κοινότητε τη κοινοτόμου γνώση. Εδώ ήθελα να γίνει κάποιο σχόλιο από την Επίτροπο. Ευχαριστώ. Ε, εντάξει, ξεπεράσαμε λιγάκι την ώρα. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ε, ισονομία μεταξύ, ισότητα μεταξύ βορρά και νότου, πλουσίων και φτωχών, ε, παλιών και καινούριων. Δεν νομίζω ότι αυτό συνέβη αυτή τη στιγμή. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank you very much. And again... Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλα τα μέλη για τις τόσο σκόπιμες και εύστοχες ερωτήσεις τους. Για τον κοινό προγραμματισμό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο παράδειγμα για το Alzheimer, ότι προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε γνώσεις από όλη την Ευρώπη και δεξιότητες από όλη την ευρωπη από πολλά κράτη-μέλη. Μιλάμε για μια πολύ καλή πιλωτική εμπειρία, όμως απαιτείται εδώ εντονότατη προσπάθεια από τους συντονιστές. Τα κράτη-μέλη διαρκώς ζητούσαν τη συνδρομή της Επιτροπής. Όμως τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι ε, θα έπρεπε και οφείλουν να δεσμευτούν και σε επίπεδο χρηματοδότησης και οικονομικών μέσων για να πετύχουμε. Για το ΙΤΕΡ. Νόμιζα ότι είχα απαντήσει και μάλιστα διεξοδικά για το ΙΤΕΡ. Σας έχω πει ποια είναι η δική μου αίσθηση γι' αυτό. Ξέρετε τι πιστεύω για τα έργα μεγάλη εμβέλεια, για τι υποδομέ που στηρίζει η Επιτροπή, αλλά μέσω ring fencing, περί χαράκωση των κομπιλίων που θα του αποδοτηθούν. Μην ξαναζήσουμε δηλαδή ότι ζήσαμε με τον Καλλιλέο και το Ίτερ. Για το πακέτο αυτό, το είχα ξεχάσει στον πρώτο γύρο ερωτήσεων, είχε τεθεί και προηγουμένω. Είναι προφανώ ευθύνη του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Όμω, να πω ότι όπω θα ξέρετε, 12 κράτη-μέλη έχουν στείλει αιτήσει στην Επιτροπή για εγκριθούν δικά τους προγράμματα και στις 14 Δεκεμβρίου ε, ενέκρινε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρόταση με για απόφαση του Συμβουλίου που θα επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία αυτών των τομέα. Ελπίζουμε ότι επί Ουγγρική Προεδρία θα εγκριθεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία οριστικώ, ίσω στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα το Μάρτιο. Πριν από αυτό, η συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου χρειάζεται και αυτή. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, από ό,τι ξέρω, ήδη έχει δηλώσει ότι στηρίζει. Στηρίζει την ταχεία λήψη απόφαση, ώστε να περάσουμε στην ε, γρήγορη υλοποίηση, διότι στην πραγματικότητα, από την οπτική γωνία τη καινοτομία, είναι ότι το κόστος ε, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες είναι 20 πλάσιο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, εδώ από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό ε, ουσιαστικά αποτελεί τεράστιο φραγμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μια αναπηρία του συστήματό μα για τι εταιρικέ σχέσει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Το είχα πει και στι αρχικέ μου απαντήσει. Εδώ θέλουμε έναν τρόπο τελείως νέο και ρηξικέλευθο για να ανανεώσουμε τον τρόπο που διασυνδέονται ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και τα προβλήματα που τώρα έχουμε αντιμετωπίσει. Χρειαζόμαστε ταχεία παροχή εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Τα προβλήματα εδώ είναι διτά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, που έχει και η κοινωνία των πολιτών μαζί μας, δηλαδή να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και βεβαίω αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, διότι η όλη έννοια ε, στηρίζεται τη στρατηγική προσέγγιση που προέκρινα και εγώ για την ε, καινοτομία και αυτό βεβαίω έχει τι ρίζε του στη στρατηγική για το 2020. Νέε πηγέ χρηματοδότηση. Ο σκοπό εδώ είναι να δημιουργήσουμε σχέση συνεργασία μεταξύ υπαρχών των προγραμμάτων και καθώς μιλούμε για τις ε, εταιρικέ αυτές σχέσεις, δεν είναι νέο μέσο. Είμαι κατά της δημιουργίας, της τέσπισης νέων μέσων, που λειτουργούν πολλές φορές ως αυτός σκοπός. Όχι. Ε, εδώ ε, εξετάζουμε όλα τα εργαλεία και τα μέσα που ήδη διαθέτουμε και είναι πολλά, σας διαβεβαιώ. Δεν χρειάζονται νέα. Ιδίως σε μια φάση που έχουμε αποφασίσει ότι κάποια από τα ήδη υπάρχοντα θα πρέπει και να εξαλειφθούν, να τα σβήσουμε. Το να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα εργαλεία σε ένα κοινό σύνολο, μια κοινή ομπρέλα όπως λέμε συχνά, σε ένα στρατηγικό πλαίσιο και σε μια κοινή κατεύθυνση βάσει των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων καινοτομία μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε το χάσμα που υπάρχει και να εξεύρουμε σφαιρικές λύσεις, πανευρωπαϊκές, για να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς προκλήσεις. Η πιλωτική εταιρική σχέση ξεκίνησε για την ενεργό ε, γύρανση, την ε, υγιή γύρανση. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εξαντλήσει τους προπολογισμούς όλων των κρατών μελών και παγκοσμίω όλες τις χώρες. Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους μόλις ολοκληρώθηκαν ε, στην πιλωτική αυτή εταιρική σχέση, αλλά πρέπει να πω ότι ε, Τελικώ χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο αποφάσισε να στηρίξει την εταιρική αυτή σχέση. Ελπίζουμε ότι παρομοίω θα λάβουμε δέσμευση από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και την ερχόμενη Πέμπτη για να στηρίξουν το σχέδιο αυτό. Για την αποτίμηση του 7ου προγράμματο πλαισίου. Μάθαμε πολλά. Μάθαμε πολλά από την διαδικασία αξιολόγηση που έγινε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων, όπου προέδρευε ο κ. Σαβενμπερκ. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε επίσημη απάντηση, απάντηση στην οποία θα φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε και μια σειρά από απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσατε. Ερωτήσει για την αξία, την προστιθέμενη αξία, του αριθμού του 21%. Δεν ξέρω πού τους βρήκατε του αριθμού αυτού. Ίσως μπορούσε ο βουλευτής που το έθεσε να μου το εξηγήσει στο τέλο. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι όπω το βλέπω εγώ τουλάχιστον η έρευνα και η καινοτομία στη χρηματοδότησή του ε, πρέπει να γίνουν αντικείμενο επενδύσεων, ώστε να προσφέρουν προσταθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που η δημιουργία του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου είναι πολύ σημαντική ως το 2004. Πρέπει αυτό να το πετύχουμε ως το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε κατακαιρματισμό των προσπαθειών. Δεν ε, θέλουμε επανάληψη των προσπαθειών. Το βλέπουμε αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αν τη δούμε συνολικά. Ε, και αν δούμε τους ερευνητές, θέμα που έθεσε νομίζω ένα από τους τελευταίους ομιλητές, νομίζω κύριο Έλλες, ε, μίλησε για τις ε, online αιτήσει. Ήρθαν πέρσι και μου υπέβαλαν αιτήσει επίσημες. Δεν μπορώ... Δεν μπόρεσα παρά να του δείξω ένα κουμπαρά που έχω πάνω στο γραφείο με μερικά νομίσματα μέσα. Και να του πω ότι υπάρχει ένα μικρό τμήμα μερίδιο ερευνητών που πραγματικά είναι σε απόλυτη. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι με πρέπει να περάσουν, με τι διοικητικέ διαδικασίε και τι αιτήσει που υποβάλλουν για χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια για τα ερευνητικά του προγράμματα. Λοιπόν, μιλήσαμε για την απλούστευση. Όπω είπε η κυρία Αντρίσεν, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάμε για την απλούστευση και να τη χρησιμοποιούμε ω όρο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι ενέργειε αναλαμβάνουμε και τι κάνουμε στην πράξη όσα προβλέπει η ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για την απλούστευση, σε ένα βαθμό είχαμε την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε και στην πράξη. Και αυτό μας επέτρεψε να έχουμε πολύ περισσότερο και πιο φιλόδοξη απλούστευση και τέτοια μέτρα. Αυτό βεβαίω είναι κάτι που το εξετάζουν ακόμα το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τώρα, ο κίνδυνο να έχουμε σφάλματα είναι κάτι που το συζητάμε ακόμη και στην, στην Επιτροπή στο επίπεδο τη ε, Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών επίση στο Κοινοβούλιο. Εκεί έχουμε ήδη συζητήσει με την κυρία, με την πρόεδρό σα, όταν ε, ενώπιον τη Επιτροπή αυτή είχα παρουσιαστεί για την απαλλαγή, την τελευταία απαλλαγή. Η συζήτηση δεν έχει ακόμη κλείσει. Όμω είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να υπάρχει πραγματική απλούστευση. Αληθινή. Όχι απλώ να τη συζητάμε την απλούστευση. Να σα δώσω έναν αριθμό. Τον είχα δώσει και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Εάν θέλουμε να πετύχουμε το 2%, το στόχο του 2%, αυτό σημαίνει επιπλέον 5.200 ε, κροάσεις ελέγχους. Δηλαδή, ανθρώπινοι πόροι, το πόσο θα πρέπει να κυνηγήσουμε και για τα μικρότερα ποσά και να είμαστε εξονυχιστικοί στον έλεγχό μας. Όλα αυτά ε, απαιτούν όχι έλεγχο μόνο των μεγαλύτερων εταιριών, των μεγαλύτερων εταίρων, ενδιαφερομένων μάλλον, όλων. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η δαπάνη κονδυλίων ευρωπαϊκών στον τομέα αυτό σωστά γίνεται για το σκοπό που αρχικά είχε οριστεί και ότι μπορεί να ελέγχεται στο τέλος της διαδικασίας και από την Επιτροπή και από το Ελληνικό Συνέδριο. Για την εκπαίδευση το έθεσε η κυρία Μαντουρέλ το θέμα της ε, κινητικότητας. Είναι πολύ σημαντική η κινητικότητα. Είναι ένας τομέας όπου η Επιτροπή και εγώ η ίδια ε, εργαζόμαστε σκληρά για να πετύχουμε αποτελέσματα. Ε, είναι ένας τομέας όπου έχουμε συνεχώς διαρροές, ε, αποστράγγιξη αποστράκηση συγγνώμη, από το πνευματικό μας κεφάλαιο, τους ερευνητέ που φεύγουν, είναι πολύ δύσκολο να του φέρουμε πίσω. Ακόμη και αυτοί που θέλουν ε, να συνδυάσουν την οικογενειακή του ζωή με τον επαγγελματικό του βίο, δεν έχουν αρκετά καλές συνθήκες εργασίας για να το καταφέρουν. Αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο τους ερευνητέ. αφορά γενικώ τι γυναίκε ερευνητές. Λοιπόν, εγώ και οι υπόλοιποι επιτροποί προσπαθούμε σκληρά να πετύχουμε πραγματική κινητικότητα, να θέσουμε σε εφαρμογή λύσεις. Λύσεις για να μην υπάρχουν πλέον διαρροές. Για την ε, βασική λοιπόν ε, εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες είναι ένα θέμα που πρέπει να το επιδιώξουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει μόνο να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τουλάχιστον και να υποδείξουμε τις δυσκολίες, τις ελλείψεις, αυτού του είδους της ε, εκπαίδευσης, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πω, αλλά αν δούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρομοίως, έχουν τις ίδιες δυσκολίες με αυτού του είδους την εκπαίδευση. Από την άλλη, εάν δούμε ανατολικά προς την Κίνα, οι επενδύσεις, οι κολοσιαίες επενδύσεις που γίνονται σε αυτόν τον χώρο, Νομίζω ότι μπορεί πολλά να μας διδάξει. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και οι ευρωβουλευτέ που έχουν επαφέ με του πολίτε πρέπει να επηρεάσουν τοπικέ και περιφερειακές κυβερνήσει ώστε να γίνουν επενδύσει. Όταν ζούμε στιγμές λιτότητας σε όλα τα κράτη-μέλη, νομίζω καλό είναι να σκεφτούμε ποια κράτη-μέλη κάνουμε τις πιο άγριες περικοπές στους προπολογισμού τους, αλλά κατάφεραν και να διατηρήσουν ή σε κάποιες περιπτώσεις να αυξήσουν τα επίπεδα δαπάνη στην έρευνα την καινοτομία και την επιστήμη. Πάντοτε ε, δίνω ως παράδειγμα την Φιλανδία. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχαν τεράστιες δυσκολίες. Οικονομικές δυσκολίες. Όμως η κυβέρνηση έλαβε τότε μια απόφαση. Επένδυσε σε στρατηγικούς τομείς, δηλαδή την έρευνα και την εκπαίδευση. Αυτό τώρα τους δίνει καρπούς. Εάν κοιτάξουμε τα κρατη μέλη προς δυσμάς, πρέπει να πω ότι παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο πληθυσμός τους, 12,5% αύξηση προβλέφθηκε στον προπολογισμό για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία και τα σχετικά προγράμματα. Αυτά είναι Αυτές τις προσπάθειες θέλουμε να δούμε να καταβάλουν τα κάτι μελη Για την επισητιστική ασφάλεια. Εδώ μιλάμε για έναν τομέα όπου εάν δούμε τις εταιρικέ σχέσεις καινοτομία τη Ευρώπη και τι μεγάλε προκλήσει για την κοινωνία των πολιτών, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επιστημιστική ασφάλεια. Εγώ είμαι γεμάτη εμπιστοσύνη ότι το Συμβούλιο, όπω και το Ευρωκοινοβούλιο, θα καταλάβουν ότι στην πιλωτική εταιρική σχέση τη Ευρώπη πραγματικά καταφέρνουμε ήδη να πετύχουμε τα πρώτα μα αποτελέσματα και αυτό με τρόπο θετικό, με τρόπο ικανοποιητικό. Αυτό ελπίζω λοιπόν να γίνει και με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ εταιρικέ σχέσει. Η βιώσιμη γεωργία είναι μία από τι υποψήφιε για αυτέ τι ευρωπαϊκέ εταιρικέ σχέσει. Ακριβώ για τον λόγο ότι η επισητιστική ασφάλεια είναι τόσο ζωτική σημασία. Παγκοσμίω πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αυτή την, πρόκληση. Και για συγκεκριμένες ε, προκηρύξεις διαγωνισμών για τον τομέα της επιστηστικής ασφάλειας που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Ιούλιο για το πρόγραμμα το 2012. Εκεί ξέρουμε ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη απόκριση. Για τα εθνικά συστήματα επαφής και το σύστημα αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι τα εθνικά σημεία επαφής ε, επιτρέπουν στους ερευνητές, τα πανεπιστήμια, τις τοπικές κυβερνήσεις των κρατών να λάβουν πληροφορίες, πληροφορίες για το πρόγραμμα πλαίσιο. Δέχομαι απολύτως τις επικρίσεις βεβαίως, τα επικριτικά σχόλια για το διοικητικό άχθος και για το πώς οι ερευνητές και οι ενδιαφερόμενοι θα προτιμούσαν να απευθύνονται αλλού παρά να πρέπει να περάσουν από όλο το διοικητικό άκθο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθεί χρηματοδότηση για την ε, καινοτομία και την ε, ε, γνώση. Εδώ, όταν ετοιμαζόμουν για την ακρόασή μου στο Ευρωκοινοβούλιο στην Επιτροπή Ήτρε, ανακάλυψα με μεγάλη μου έκπληξη ότι στα κάτι μέλη που γνώριζα καλύτερα την κατάστασή του υπήρχε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία είχε ιδρυθεί για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνον για να εξηγεί τα προγράμματα πλαίσιο στου ενδιαφερομένου. Όχι μόνο σε ένα κράτο μέλο, αλλά και σε άλλα υπήρχαν τέτοιε καταστάσει. Αυτό αποδεικνύει, δεν χρειάζεται κι άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ότι και μεγάλο άχθο υπάρχει και υπερβολικό το άχθο αυτό είναι και πρέπει να ε, πάυσουν, να εξαλειφθούν τα απαγορευτικά και να τα ξεχάσουμε τελείως, να αφήσουμε πίσω μας. Για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, νωρίτερα αυτό το μήνα, είχαμε μια πρώτη απόκριση. Εδώ θα επανέλθω και στην Επιτροπή Ήτρα για να παρουσιάσω αυτή μας την απάντηση. Το πρόγραμμα ITER. Ξανά το ITER, το Γαλιλαίο, όλα αυτά τα μεγάλες εμβέλειας προγράμματα που προβλέπουν μεγάλε υποδομέ και δεν πήγαν καλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν θα πρέπει να μα φέρουν στην ίδια θέση. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να λένε όταν αυξάνονται τα κονδύλια, όταν ε, τελειώνουν αυτά που του δίνει ο προπολογισμό να πηγαίνουν πάλι στην Επιτροπή και να ζητάνε. Όχι, δεν είναι δίκαιο ούτε για του επιστήμονε και του ερευνητέ. Ε, μπορούν άλλωστε να ισχυριστούν ότι ε, εάν. Μάλλον δεν είναι δίκαιο ε, για επειδή εξαντλήθηκαν τα κονδύλια του εθνικού προπολογισμού, να πηγαίνουμε και να τα παίρνουμε αυτά από άλλα προγράμματα ή από άλλου τομεί. Πρέπει να υπάρχει εδώ το λεγόμενο ring fencing, αυτή η περιχαράκωση που λέγαμε και πριν, ώστε να ξέρουμε τι αποδίδεται πού για την διαστημική πολιτική. Αυτό είναι κάτι που το διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Εδώ δεν μπορούσε να υπάρχει ένας επίτροπος ε, ε, πιο αφοσιωμένο στη διαστημική πολιτική και την επιχειρηματικότητα από ότι ο Επίτροπο Σταγιάννη, ο Αντιπρόεδρο Σταγιάννη. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλα τα ζητήματα τη έρευνα και τη καινοτομία. Για τον συντονισμό των κρατών μελών ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πώς θα έχουμε εναρμονισμένη χρηματοδότηση, συντονισμένη χρηματοδότηση καλύτερα. Εδώ μην ξεχνάμε και το άρθρο 169 το παλιό 169 που έχει γίνει 185 τώρα. Εδώ ορίζεται κοινό προγραμματισμό. Οι πρωτοβουλίε αυτέ ανταποκρίνονται στο 10%, το 10% του 7ου πλαισίου. Πρώτα απ' όλα, όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει σαφή ανάγκη συντονισμού και έπειτα χωρί να δαπανίσουμε περισσότερα κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο συντονισμό πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει του ε, ε, αυστηρού κανόνε ε, που ανάγονται σε μια δεκαετία νωρίτερα Συντάξει, επιδόματα, δυσκολεύουν την κινητικότητα των ερευνητών, ε, επικαλύψεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο και περιορισμούς μεταξύ των κρατών. Εδώ υπάρχουν διαφορετικά εθνικά προγράμματα που καλό θα ήταν να συνενωθούν σε ένα ευρωπαϊκό σύνολο, μια κοινή ομπρέλα, αλλά όχι ένα ενιαίο μόνο πρόγραμμα. Εδώ θέλουμε να συνδυάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και να στηρίξουμε και την πολιτιστική ποικιλότητα που υπάρχει ούτως ή άλλως στο επίπεδο τη έρευνας και γενικότερα στα ακαδημαϊκά το Eurostar είναι ένα χαρακτηριστικό, το Eurostar είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ε, που ε, ε, βάσει του άρθρου 185 πρόσφερε κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπόρεσε να διασυνδέσει εθνικά προγράμματα όπως το Eureka, το Εύρικα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι λίγο πολύ απάντησα σε όλα. Τα νέα κατημέλη. Τα νέα κατημέλη Πάντοτε μα έλεγαν ότι δυσκολευόμαστε να πετύχουμε την αριστεία. Ιδίω αν το δούμε αυτό από την άποψη τη ευρωπαϊκή έρευνα και τι δωρεέ που δίνονται, τι επιδοτήσει. Ε, είναι πολύτιμε, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αλλού εξυπηρετούν του σκοπού του. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι εκείνη θέτει τι προδιαγραφέ τη αριστεία για όλου του ερευνητέ, παγκοσμίω. Τα νέα λοιπόν πολύ συχνά έρχονται και μου λένε κοιτάξτε δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πετύχουμε το είδος αριστείας που απαιτείται. Τι λέω λοιπόν εγώ τότε, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η αριστεία να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί να το συνδυάσουμε με τις υποδομές τους. Ερευνητές έχουν, επιστήμονες έχουν, αλλά έχουν δυσκολία οι περισσότεροι από αυτούς να μπορέσουν να τους κρατήσουν στη χώρα, να τους προσφέρουν υποδομές και εγκαταστάσεις που να τους ενθαρρύνουν να μείνουν και να ενθαρρύνουν και άλλους να έρθουν τους ε, κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές να εργαστούν εκεί. Πρέπει λοιπόν αυτό να καλλιεργηθεί. Αυτό το επίπεδο αριστείας θέλουμε να αναπτυχθεί. Τέλος, να πω ότι υπολογίζω στη στήριξή σα και τη δική σα τη δέσμευση και αφοσίωση. Νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι η ερευνητική πολιτική ή μια άλλη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηριχθούν. Όχι, εγώ δεν τα σκέφτομαι τα πράγματα έτσι. Η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να γίνονται αντιληπτέ ω μέρο των υπόλοιπων πολιτικών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το προωθήσει αυτό, δηλαδή να το βλέπουμε από την άποψη των ε, επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων σε όλου του τομεί. Να σκεφτούμε πώ η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να στηρίξουν και να συνεισφέρουν σε όλε τι πολιτικέ τη Ένωση. Με άλλα λόγια, το να μετακινηθεί, το να αλλάξει η γενική διεύθυνση από το να γίνει ε, μια διεύθυνση που προσφέρει απλώ ε, κίνητρα τους ερευνητές, ε, να γίνει μια γενική διεύθυνση που δίνει και πολιτικές κατευθύνσεις, που στηρίζει τις πολιτικές άλλων γενικών διευθύνσεων. Θα πρέπει οι Επίτροποι όλοι μαζί και εσείς να στηρίξουμε την προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτών των διεθνών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και των στόχων που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Στατική του 2020. Ε, Ευχαριστώ. Ιδίω όσον αφορά την νοοτροπία ή μάλλον την αλλαγή ε, νοοτροπίας ε, σχετικά με τις ε, διοικητικές μεθόδους. Ευχαριστώ, αλλά η Έλγα Τρίπελ είχε ακόμη μία σύντομη ερώτηση. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα, διότι θα ήθελα να ξέρω πόσο η δομή αυτή του one-stop shop θα λειτουργήσει στην καθημερινή ζωή. Δεν το έχω αντιληφθεί και θα ήθελα να μπορέσω να το καταλάβω. Καταρχήν, είτε μιλάτε για περιφέρειες ή για κράτη-μέλη, έχετε εθνικά σημεία επαφής, τα οποία υπάρχουν για να μπορούν να ενημερώνουν, να εκπαιδεύουν, να εμπλέκουν τους ενδιαφερόμενους σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο και ε, να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει η πλαισίωση και στηρίξή τους μέσω αυτού του σημείου. Αλλά χρειάζεται ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο να περιλαμβάνει την ε, ευρωπαϊκή συμμετοχή στο EIT, το SIP και το πρόγραμμα πλαίσιο. Δηλαδή εφόσον θα υπάρχει αυτό το κοινό πρόγραμμα θα εξετάζουμε τη χρηματοδότηση όχι η βάση του τι έχουμε στο σημείο αλλά τη συνολική ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα ε, διαθέτει χρηματοδότηση έτσι με ένα σημείο εισόδου το οποίο θα είναι προφανώς στις Βρυξέλλες διότι ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα κόσμο όπου χρησιμοποιούμε συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή είτε βρίσκεστε στις Βρυξέλλες ή στη Ρήγα έχετε πρόσβαση ή ε, στην ισοσελίδα της Διευθύνσεως Έρευνας και Καινοτομίας. Έχετε τρόπους να ενημερωθείτε ε, ανα πάσα στιγμή ε, και από εκεί αλλά και μέσω των σημείων επαφής σε εθνικό επίπεδο όπου μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι εμπλεκόμενοι για όσους συμμετέχουν πρώτη φορά στη διαδικασία χρηματοδότησης και ε, ζητούν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ένα από τα κοινά σημεία εισόδου περιέχει ένα κοινό σύνολο κανόνων όπου δηλαδή εσείς κάνετε την αίτησή σας ε, είσαστε μια μικρομεσαία επιχείρηση και όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή εγγυόμαστε το 50% του προγράμματος πλαισίου που πρέπει να διοχετευτεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται κατά τη συζήτηση του MFF να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό αλλά είναι κάτι που πρέπει ακόμη να αποφασιστεί και όταν έρχεστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο μηχανισμό χρηματοδοτήσεως άπαξ και αποφασιστεί στο πρώτο σημείο επαφής ότι είστε μικρομεσαία επιχείρηση, ανεξαρτήτως από πού προσπαθείτε να χρηματοδοτηθείτε πάντοτε θεωρείστε μία μικρομεσαία επιχείρηση ενώ τώρα εάν θεωρείστε ότι είστε μία μικρομεσαία επιχείρηση και μετά διαπιστωθείτε ως πρόγραμμα πλαίσιο δεν ε, ε, ε, πρέπει να ξαναξιολογηθεί ο φάκελός σας άρα υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός του γραφειοκρατικού άχθους το οποίο πρέπει να αποφύγουμε και να απεμπλακούμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία μία βάση δεδομένων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην χρειάζεται ε, πλέον σε κάθε γενική διεύθυνση. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα χρησιμοποιούσαμε. Ναι, αλλά αυτή ήταν η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2006 τότε χαιρόμαστε που η, Επιτροπή, η Επίτροπος τουλάχιστον επωφελήθηκε της καλής μας ιδέας. Το αποτέλεσμα είναι το, το ίδιο και το αυτό. Οπότε, Τώρα παρακαλώ το Σαλβαντόρ πολύ σύντομα να χρησιμοποιήσει ό,τι η ενέργεια του έχει απομείνει κατά τρόπο ώστε στο τέλος μιας μακριάς ημέρας να ψήσει ε, τη συζήτησή μας σε αυτό το θέμα της Μερσίας διατάξεως. Πρόεδρε. Ε, νομίζω είναι αδύνατο να συνοψίσω ε, στο βαθμό της λεπτομέρειας που μας έδωσε η Επίτροπος με τις απαντήσεις της, ε, μένα μου είναι αδύνατο να συνοψίσω. Βέβαια, υπήρξαν αρκετές ε, σαφείς ιδέες που προέκυψαν, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκπονήσουμε την τελική μας ε, έκθεση. Έχει καταστεί σαφές ότι είναι ε, σημαντική η ε, πολιτική έρευνα και καινοτομία, η οποία να είναι πλήρω χρηματοδοτούμενη. Οπότε, όταν θα παίρνουμε χρηματοδοτικέ αποφάσει για θέματα που σχετίζονται με αυτούς του τομεί, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην Επιτροπή μας. Κάτι που μου έκανε εντύπωση όταν μίλησε η Επίτροπος για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και την προετοιμασία για το 8ο. Είπε ότι θα πρέπει να καλύπτει όλη την λυσίδα από την ε, έρευνα στην αγορά. Και νομίζω ότι αυτό όντω είναι σωστό και συνάδει και με τη στρατηγική 2020 και τους στόχους για την ανάπτυξη, την, ε, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την Επίτροπο. Eh, Επίσης, νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται ένα στρατηγικό πλαίσιο, ε, κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη. Είναι σαφές, ε, δόθηκαν πολλά παραδείγματα, ε, ότι το 80% όχι μόνο γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 80% της έρευνας, αλλά ακόμη και σε κοντινές χώρες βλέπουμε άμεσο ανταγωνισμό από μεγάλους ε, ε, κολοσσούς ε, βιομηχανικούς όπως η Κίνα που λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της το θέμα της έρευνας και θα πρέπει λοιπόν και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε για το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν έχουμε ακόμη το απαραίτητο χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για να προχωρήσουμε στον τομέα όπου χρειάζεται περισσότερο. Πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε να έχουμε προστιθέμενη αξία. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι κατακαιρματισμός και επικαλύψεις. Χρειάζεται καλός συντονισμός με, τις, ε, με τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα και αυτό και νομίζω ότι έτυχε μεγάλη υποστήριξη στη συζήτηση, θα μπορούσε να, προσθέσει, να φέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ότι όλες οι υπόλοιπε ε, συμφωνίες για την, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα, ε, ήταν αρκετά πιστικά τα επιχειρήματα που ακούσαμε, οπότε δεν θα πρέπει απλώς να δίδουμε ενίσχυση για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για τα εθνικά που μπορούν να ε, πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου. Προ το παρόν δεν υπάρχει ε, δυνατότητα για σύνδεση όλων αυτών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει όντω να το δούμε σοβαρά. Γιατί μόνο ένα από τα τρία ερευνητικά προγράμματα που ζητά χρηματοδότηση γίνεται δεκτό. σω γιατί είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία. Αλλά σίγουρα αυτόν τον αριθμό θα πρέπει να τον αυξήσουμε. Η Επίτροπο επίση, στο τελικό του σχόλιο, είπε ότι είναι δυνατό κάποια από τα χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα και την κοινοτομία να εξαφανιστούν ότι είναι πιθανό αυτό ή να εξαφανιστούν ή να αλλάξουν. Τέτοιου είδους ε, δηλώσεις ε, δυσκολεύουν τη ζωή των εισηγητών πρέπει να πω γιατί δίνει, ε, εισάγουν μια μεγαλύτερη ανασφάλεια όταν θα εκπονήσουμε την τελική εκδοχή του κειμένου μας και εμείς μιλήσαμε για απλούστευση και νομίζω ότι υπήρξε στήριξη από την Επιτροπή ότι η απλούστευση, η απλοποίηση είναι κάτι που πρέπει να εισαχθεί στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο δηλαδή, και, στις, και στον δημοσιονομικό κανονισμό. Δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς, εάν υπήρχε περισσότερη απλοποίηση, η ζωή των ερευνητών θα γινόταν πιο εύκολη. Καθώς επίσης και η ζωή των ελεγκτών. Αν, δείτε, αν το δείτε αυτό από την πλευρά του κοινού στρατηγικού πλαισίου, ε, αυτό είναι λογικό και αυτό θα φαίνεται στην τελική μας έκθεση. Επίσης, χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια και καλύτερο, πιο σταθερό πλαίσιο για, την, ε, για, την, ε, για τα προγράμματα τα ερευνητικά, για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα όπω το ΙΤΕΡ, το συζητήσαμε αρκετά και νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ω προ αυτό και ο Γαλιλαίο επίση και το πρόγραμμα GMS. Είπαμε ότι θα χρειαστεί ίσως περιχαράκωση της ε, χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αποκλειστικά για αυτά τα μεγάλα προγράμματα. Και θεωρώ ότι αυτή είναι καλή ιδέα, γιατί αν υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση, αν υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, τότε είναι πιο εύκολο να υπάρξει δημόσια και ιδιωτική επένδυση. Μέχρι στιγμή δεν τα έχουμε καταφέρει στο Γαλιλαίο ω προς αυτό. Υπάρχουν ακόμη βέβαια κάποιες αμφιβολίες για το EIT, για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτό ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα που θα εξαφανιστεί, γιατί αυτό είναι ένα πρόγραμμα μέσω μακροπρόθεσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ελπίσουμε ότι θα ε, συνεχιστεί και η τρίτη φάση, ε, γιατί αλλιώς θα έχει μεγάλες ε, οικονομικές επιπτώσεις. Στο μέλλον νομίζω ότι θα χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν. Και τέλος, αριστεία. Νομίζω ότι η αριστεία, όπως έχουν τα πράγματα, είναι περισσότερο στόχος παρά κριτήριο για απονομή κονδυλίων. Νομίζω ότι η αριστεία μπορεί να επιτευχθεί μέσω του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Γιατί αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές. Έχουμε εξαιρετη, εξαιρετο τομέα έρευνας. Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη ε, απόδοση των κονδυλίων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επαναλάβω την, ε, τις ευχαριστίες μου προς την Επίτροπο και να εκφράσω την ε, χαρά μου για το υψηλό επίπεδο συζήτησης που έγινε σήμερα. Ε, ξέρω ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομεριών στην έκθεσή μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τον τρόπο με τον οποίο απάντησε τις, ε, στα ερωτήματα που της θέθηκαν. Επίσης, να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο για τον εξαιρετικό τρόπο που προείδρευσε τη σημερινή συζήτηση. Φεύγω λοιπόν πολύ ικανοποιημένο με το όσα πετύχαμε από τη σημερινή συνεδρίαση. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Κλείσαμε και το σημείο 8 τη ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ και πάλι πολύ την Επίτροπο που έκατσε λίγο παραπάνω μαζί μας από ό,τι είχε σχεδιάσει. Αυτό που προκύπτει από το τελευταίο σημείο είναι ότι για τη δομή ε, θα πρέπει να καθορίσουμε την τελική εκδοχή των, ε, της έκθεσής μας για την τελική δομή των προγραμμάτων αυτών. Ίσως να πρέπει να βάλουμε ένα γενικό τίτλο «Μεγάλα προγράμματα». Νομίζω ότι αυτή η, πρώτα, η πρόταση είναι αρκετά ελκυστική και νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Να ευχαριστήσω για αυτή την ε, ε, σημαντική συζήτηση που έγινε, ε, τη γραμματεία, γιατί πραγματικά χρειάστηκε πολλή προετοιμασία για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή γιατί πραγματικά έκανε μεγάλη μάχη γιατί έπρεπε να κάνει την εισαγωγή, να κάνει την περίληψη στο τέλος. Όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν ότι υπάρχουν ε, διάφορες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εκθέσεων. Είναι πάντα θέμα συγκέντρωσης να παρακολουθεί κανείς τόσο επισταμένα όπως το έκανε σήμερα ο Σαλβαδόρ. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση λοιπόν για όλα τα σημεία της ημερησίας διάταξης πρέπει να πω ότι αναφέρθηκε τόσο συχνά η ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως νέος εταίρος για νέα ε, ε, μέσα χρηματοδότησης. Αν αναφέρεται τόσο, αν κάθε φορά που ακούγαμε το όνομα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας Επενδύσεων είχαμε 5 ευρώ, θα είχαμε σίγουρα τον, τον πρώτο κορβανά έτοιμο για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Mm-hmm. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, καλό σας απόγευμα. Πέρα συνεδρία σας. Yeah. Yeah. Yeah.